Καλημέρα σε όλους. Σας έχουμε διανύμει μια αναθεωρημένη μερίσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις με τη νέα αυτή μερίσια διάταξη μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται. Στη συνάντηση τώρα των συντονιστών που έλαβε χώρα στις 30 Αυγούστου αποφασίστηκε να ανοίξει μια χρονική περίοδος για κατάθεση τροπολογιών για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την πράξη της Γενέβης για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις. Εδώ ακολουθούμε μια διαδικασία σύμφωνης γνώμης καθώς επίσης και όσον αφορά τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην πράξη αυτή. Εδώ πέρα ακολουθείται η συνήθι νομοθετική διαδικασία. Επομένω, δεν πρόκειται να υπάρξει συντάκτη γνωμοδότηση στην Επιτροπή μα και δεν πρόκειται να συνταχθεί σχέδιο γνωμοδότηση. Οι τροπολογίε οι οποίε θα εγκριθούν στην Επιτροπή μα θα παρουσιαστούν σε μία γνωμοδότηση εξ ονόματο του Προέδρου μόνο. Επομένως σας προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα και για τις δύο προτάσεις Επιτροπής. Η καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση τροπολογιών στην ΕΜΒΗ 25 Οκτωβρίου, ως συνήθως μέχρι τις 11 το πρωί, θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 26-27 Νοεμβρίου και κατά πάση πιθανότητα στην Επιτροπή Γιούρη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τον Ιανουάριο. Δεύτερη ανακοίνωση κοινή συνάντηση των Επιτροπών Άγκρι Agri-NVK3 και Ιτρέ όσον αφορά τα δάση. Μετά από πρωτοβουλία της Επιτροπής Γεωργικών Υποθέσεων, αποφασίστηκε μία κοινή συνάντηση των Επιτροπών Γεωργίας Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας για την στρατηγική τη δασική, δασική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνάντηση αυτά τη χώρα στο Στρασβούργο στις 14 Ιανουαρίου. Στόχος είναι να γίνει αλλαγή απόψεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζουμε με την παρουσία του Επιτρόπου Χόγκαν σε σχέση πάντα με την ε, ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση. Κατόπιν έχουν γίνει κάποιες αλλαγές όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των δικών μας συναντήσεων. Η απογευματινή ε, συνάντηση προβλεπόταν για τις 8 Νοεμβρίου, δεν θα λάβει χώρα, θα συνεδριάσουμε εκείνη τη μέρα μόνο το πρωί και θα σας ε, διανεμηθούν εν ευθέτω χρόνο οι ημερήσεις διατάξεις. 21 γλώσσες προβλέπονται για σήμερα όσον αφορά την διερμηνία και τα έγγραφα έχουν διανεμηθεί ηλεκτρονικά και βέβαια η συνεδρίασή μας μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Τώρα συστάσεις των συντονιστών από τις συνεδρίες της 10ης Οκτωβρίου. Οι συστάσεις αυτές σας έχουν διανεμηθεί ηλεκτρονικά και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Επίσης, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, τα πρακτικά των συνεδριάσεων τη 9 η και 10 η Ιουλίου, καθώς επίση και της 13 η Σεπτεμβρίου, που και αυτά σας έχουν διανεμηθεί, θα θεωρηθούν και αυτά ότι έχουν εγκριθεί. Α περάσουμε τώρα στο πρώτο θέμα συζήτηση, στην σημερινή ημερήσια διάταξη. Έχουμε δύο αντιρρήσει, όσον αφορά τον γενικά, γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο. Δεν πρόκειται να σας διαβάσω όλο τον τίτλο του σημείου αυτού, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές ποικιλίε αραβόσιτου. Ο τίτλος εδώ πέρα είναι πολύ μακροσκελής. Σας προτείνω να πάρετε το λόγο, να μας παρουσιάσετε τις αντιρρήσεις αυτές και θα ακούσουμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ας ξεκινήσουμε με τους συνεισηγητές. Ο κύριος Στές πρώτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώ δεν είναι πολλοί συνάδελφοι σήμερα εδώ. Μου προκαλεί εντύπωση αυτό γιατί το, το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι πρώτη φορά που ασχολούμεθα με το ζήτημα αυτό. Σε προηγούμενε αντιρρήσεις ήταν περισσότεροι οι συνάδελφοι και ήταν και πιο έντονη η συζήτηση που ακολούθησε. Και ξέρετε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε πλειοψηφία των βουλευτών που εγκρίνουν τι αντιρρήσεις και έχουμε πολλές φορές και τα δύο τρίτα των βουλευτών στην Ολομέλεια που εγκρίνουν τελικά τις αντιρρήσεις που προτείνουμε. Σε κάθε περίπτωση η σημερινή αντίρρηση έχει να κάνει με γενετικά τροπημένους οργανισμούς που έχει προτείνει η Μονσάντο Ευρώπης και εδώ πέρα έχουμε γενετικά τροποποιημένο ραβόσιτο που συνδυάζεται με δύο, τρεις ή τέσσερις διαφορετικές ποικιλίε. Συγκεκριμένα γενετικά τροποποιημένο ραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα. Τα βλέπετε αυτά στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Αναφερόμαστε εδώ πέρα στην, στον κανονισμό του 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς έχουμε προβάλει μία αντίρρηση όσον αφορά την ανανέωση της αδειοδότησης. Είχαμε 27 επιτυχείς αντιρρήσεις στο παρελθόν, ακόμα και στο Συμβούλιο των Υπουργών. δεν καταφέρνουμε να έχουμε τέτοια πλειοψηφία σαν αυτή που είχαμε πετύχει εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλες αυτές τις παρελθούσες αντιρρήσεις. Στις 11 Σεπτεμβρίου στη Μόνιμη Επιτροπή υπήρχαν ε, τέσσερα κράτη-μέλη τα οποία ήταν κατά, 11 υπέρ και τα υπόλοιπα πήγαν. Και είχαμε και μια άλλη ψηφοφορία 13 κατά και 4 αποχές. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει εδώ πραγματικά ένα ζήτημα δημοκρατικής νομιμότητος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά δεν λαμβάνει υπόψη στην την αντίρρηση τόσο του Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου των Υπουργών. Να σα υπενθυμίσω ότι μόνο και μόνο η δική μα η Επιτροπή, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, έχει, έχει εγκρίνει Μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορθώνει Ομιλητή έχει εγκρίνει περισσότερε ενδοδοτήσει από ό,τι προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα πολλέ διαφορετικέ ποικιλίε γεντικά τροποποιημένου αραβόσιτου που προτείνονται και η ίδια Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων, η ΕΦΣΑ, έχει παραδεχθεί ότι για 14 υποενώσεις αραβοσίτου από αυτού που προτείνονται δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες επιστημονικές πληροφορίε και στοιχεία από την ίδια την Μονσάντο. Το παραδέχεται αυτό η ίδια η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Επίσης κάποιες υποενώσει που προτείνονται δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί. Έχουν πει ότι για πέντε ποικιλίε δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι δεν έχουν γίνει επιστημονικές δοκιμές. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ε, ενώσεις αραβοσίτου, γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο που είναι ανθεκτικό τόσο στο γλυφοσάτι όσο και στο γλυφοσονικό αμμόνιο. Γνωρίζουμε ότι οι ουσίες αυτές είναι καθαρά τοξικές ουσίες και ξέρετε ότι προβλέπονταν συγκεκριμένε εξαιρέσει ήδη από το 2009 όσον αφορά τι ουσίε αυτέ. Επίση, η ανθεκτικότητα στα ζυζανιοκτώνα που περιέχουν γλυφοσάτι ή γλυφοσονικό αμμόνιο είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Πρόκειται για ουσίες οι οποίες πολλές φορές στο παρελθόν έχουν απαγορευτεί, έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το οποίο προτείνεται τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με αυτά τα οποία έχουμε εγκρίνει στο παρελθόν εδώ στα πλαίσια της Επιτροπής μας, στα πλαίσια της κοινοτικής τελικά νομοθεσίας. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και σταθμά σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν εντό και εκτό Ευρώπη. Θεωρώ ότι αν εγκρίνουμε τι ουσίε αυτέ, τον γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο, θα έχουμε σε χώρες όπως το Μεξικό και η Νότιο Κορέα περισσότερη παραγωγή των ουσιών αυτών. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι λένε ότι δεν έχουν γίνει απαραίτητε δοκιμέ. δεν έχουν γίνει οι απαραίτητε επιστημονικέ μελέτε, δεν έχουν γίνει απαραίτητε μελέτε στα τροπτικά που πρέπει να είχαν γίνει και υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που λένε ότι τα στοιχεία αυτή τη στιγμή είναι ανεπαρκή σε σχέση με τι ανεπιθύμητες επιπτώσεις που θα μπορούσαν να είχαν αυτές οι ενώσεις γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου. Ακριβώς λοιπόν επειδή υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα όσον αφορά τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην ανθρώπινη υγεία αλλά και στο περιβάλλον οι ουσίες αυτές, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να προβάλλουμε την αντίρρηση αυτή. Παρ' όλα αυτά όμως, και αυτό μας προκαλεί εντύπωση, η ΕΦΣΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων, δεν έχει προβεί στην απαραίτητη δράση όσον αφορά τον έλεγχο της διάθεσης των προϊόντων αυτών στην αγορά. Γι' αυτό το λόγο και εγώ και οι υπόλοιποι συνεισηγητές, απευθυνόμενοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέμε ότι δεν τηρεί αυτή τη στιγμή του ίδιου του κανονισμού που υφίστανται όσον αφορά την προστασία τη ανθρώπινη υγεία, τη υγεία των φυτών και τη υγεία των ζώων και γενικότερα του κανονισμού που υφίστανται για την προστασία του περιβάλλοντο και τη δημόσια υγεία. Έτσι λοιπόν η αδειοδότηση αυτή η οποία ζητείται αυτή τη στιγμή για να μπορεί να εισαχθεί την κοινοτική αγορά η νέα αυτή μορφή γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου είναι κάτι το οποίο αντιτίθεται στην κοινοτική νομοθεσία. Επαναλαμβάνω, δεν έχουν γίνει δοκιμέ, δεν έχουμε τα επιστημονικά δεδομένα και κυρίω ορισμένε από τι ενώσει αυτέ αραβόσιτου δεν υπάρχουν καν, δεν έχουν δημιουργηθεί. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο τύπο του, που προτείνεται στο σημείο 6 μερίσια διάταξη, έχουμε τι ίδιε ενστάσει εδώ. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, η ΕΦΣΑ δεν έχει την παραμικρή πληροφορία. Έχει βασιστεί απλώ σε αυτά τα οποία έχει υποβάλει ως στοιχεία η Μονσάντο Ευρώπης. Και βάσει αυτών η ΕΦΣΑ μας λέει ότι ε, δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις, νέα στοιχεία τα οποία να δημιουργούν την υπόνοια ύπαρξη κινδύνου. Αν όμω δεν κάνουμε εμεί οι ίδιοι εδώ πέρα τι απαραίτητε έρευνε, τι απαραίτητε μελέτε, δεν μπορούμε πραγματικά να γνωρίζουμε αν υφίσταται ή όχι κίνδυνο και απλώ επαφιόμαστε σε αυτά τα οποία μα λέει εν προκειμένου η Μονσάντο. Και στη δεύτερη αυτή περίπτωση έχουμε το ζήτημα της γλυφοσάτης καθώς επίσης και του γλυφοσονικού αμμονίου γίνεται αναφορά εδώ πέρα στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, τι Φιλιππίνες, την Ιαπωνία, την Νότια Αφρική και την Ουρουάη. Χώρε δηλαδή στις οποίε έχουν χρησιμοποιηθεί οι ουσίε αυτέ. Ολοκληρώνοντα λοιπόν κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει να σα πω ότι είχαμε άτυπε συναντήσει με νομομαθείς εμπειρογνώμονε που γνωρίζουν το τομέα αυτό τη κοινοτική νομοθεσία και οι οποίοι ίδιοι μα είπαν ότι η πρόταση αυτή τη ευρωπαϊκή επιτροπή βρήθη προβλημάτων. Πρέπει λοιπόν να είμαι απόλυτα ειλικρινή απευθυνόμενο εκπροσώπου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέγοντά του ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να μπορούν να δικαιολογούν εδώ πέρα τι υπονεώσει 34 και 17. Πώς μπορεί ποτέ να δοθεί για τις ενώσεις αυτές δεκαετής άδεια διάθεση στην αγορά χωρίς να έχει ακολουθηθεί ιδέουσα διαδικασία προέγκρισης, όπως ακριβώς προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία. Πώς μπορούμε να εγκρίνουμε για 10 χρόνια τις συγκεκριμένες υποενώσεις αραβοσίτου. Πώς γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε μια τέτοια πράξη. Αυτή είναι η ερώτηση που υπευθύνω σε προσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσβλέπω επίσης απόψη των υπολοιπών συναδέλφων, καθώς επίσης και στην ψηφοφορία που θα έχουμε στις 10. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Εύη. Χίλια ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ τον συνάδελφο Στάε που μας παρουσίασε τις δύο αυτές αντιρρήσεις. Δύο αντιρρήσει που μας βρίσκουν συσπηρωμένους, απευθυνόμενοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητώντα τη να μην αδειοδοτήσει για την ευρωπαϊκή αγορά αυτούς τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Για μία ακόμη φορά βλέπουμε ότι αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των γενετικά αυτών τροποποιημένων οργανισμών και βλέπουμε ότι η Επιτροπή Juncker τελικά αυτή η οποία έχει αδειοδοτήσει τους περισσότερους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς σε σχέση με τις υπόλοιπε ευρωπαϊκές επιτροπές, δηλαδή τις δύο θητείες του Πρόντι και του Μπαρόζο. Πραγματικά είναι πολύ διάζουσα η κατάσταση αυτή και για μία ακόμη φορά βρισκόμαστε υποχρεωμένοι να προτείνουμε αντιρρήσεις, ενστάσεις, οι οποίες είναι απόλυτα τεκμηριωμένες. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η διαδικασία αυτή είναι καθαρά αντιδημοκρατική και δεν είμαι η μόνη που το λέω αυτό, ότι οι υπόλοιποι συνάδελφοι ο ίδιος ο πρόεδρος Γιούγκε πριν από πέντε χρόνια μας είπε ότι υφίστανται αυτές οι αντιδημοκρατικές ή αν θέλετε μη δημοκρατικά νομοποιημένες διαδικασίες και ότι θα έκανε κάτι γι' αυτό, αλλά συνεχεία δεν έκανε τίποτα. Μολονότι στο παρελθόν έχει απορρίψει σχετικέ προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αλλάξει εντελώ η τακτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί για μία ακόμα φορά βρισκόμαστε απέναντι σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση. Το τονίζω για μία ακόμη φορά, το είπε και ο συνάδελφο Στάες πριν από λίγο. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων δεν έχει χρησιμοποιήσει τα απαραίτητα επιστημονικά στοιχεία. Υπάρχουν πάρα πολλά επιστημονικά κενά και από ό,τι φαίνεται για μία ακόμα φορά και στο Συμβούλιο δεν υπήρχε ειδική πλειοψηφία προκειμένου να εγκριθούν από, την, από το Συμβούλιο με αποτέλεσμα τελικά να ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει την τελική απόφαση. Θεωρώ ότι αυτό είναι απαράδεκτο, ιδίω απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή ποτέ να ιδιοδοτούμε στην αγορά τέτοιες ουσίες οι οποίες μπορούν να έχουν τεράστιους κινδύνους. Ξέρετε μάλιστα ότι υπάρχει και μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία των πολιτών, όπως αυτή που έχει τίτλο Stop Glyphosate. Σταματήστε, τη χρήση της γλυφοσάτης περιμέναμε ότι ιδίω μετά από αυτό θα υπήρχε πραγματικά μία εσπευσμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να αλλάξει η κοινοτική νομοθεσία που έχει να κάνει με την ασφάλεια των τροφίμων. Ελπίζω ότι θα ασχοληθεί η τρέχουσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το ζήτημα αυτό και ότι θα το αναθέσει στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει η πιο υψηλή διαφάνεια σε σχέση με τη χρήση επιστημονικών δεδομένων και σε σχέση με την έγκριση των επιστημονικών αυτών δεδομένων. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή φύστανται πάρα πολλά κενά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της πολύ σοβαρά τετήματα των Ευρωπαίων πολιτών και εν γέννη δεν θα πρέπει να διοθοτήσει στην ευρωπαϊκή αγορά τι ουσίε αυτέ χρησιμοποιώντα τι μεθόδου του παρελθόντος. Τι μεθόδου αυτέ, τι προβληματικέ, δεν μπορούμε πλέον να τι δεχθούμε. Θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση. Από προσωπική πλευρά θα ήθελα να συνεχίσω να αντιτάσσομαι στην αδειοδότηση τέτοιων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, ακριβώς επειδή βλέπουμε ότι οι γενετικά αυτοί οι τροποποιημένοι οργανισμοί ουσιαστικά χρησιμοποιούνται για να χρησιμοποιείται μια πρόφαση μάλλον ότι μέσω των γεννητικών αυτών τροποποιημένων οργανισμών θα λύσουμε το θέμα του υποσυτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι μια πρόφαση μόνο. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι καλλιεργούνται οι, γενετικοί, οι γενετικά οργανισμοί με μεθόδους γεωργικές οι οποίες δεν είναι βιώσιμες, οι οποίες είναι πολύ επικίνδυνες για το περιβάλλον ακριβώς επειδή χρησιμοποιούν πάρα πολλές χημικές ουσίες και ουσιαστικά προωθούν την εντατική καλλιέργεια καθώς επίσης και την εντατική κτηνοτροφία. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και εδώ στην Ευρώπη έχουμε όλο και μεγαλύτερες ποσότητες γενετικά τροποποιημένων ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή κτηνοτροφία για να παράξουμε τελικά κρέας χαμηλής τιμής, χαμηλής ποιότητος προκειμένου να κερδοφορήσουν περισσότεροι οι πλούσιοι, θέλετε, του κόσμου αυτού ή οι πλούσιοι της Ευρώπης θεωρώ ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με το παράδεκτο αυτό μοντέλο. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι αυξάνονται πάρα πολύ τα επικίνδυνα υπολείμματα της βιομηχανικής αυτής γεωγραφίας και εκνοτροφίας. Θα πρέπει και αυτό να το έχουμε υπόψη μας και να αλλάξουμε εντελώς το μοντέλο καλλιέργειας το οποίο χρησιμοποιούμε. Δεν βλέπω άλλους ε, συνεισηγητές. Η κυρία Μαγιούσο. Υπάρχουν ε, δύο διαφωνίες ε, σχετικά με την ε, έκδοση άδεια και μια επανέκδοση άδεια σχετικά με σχετικά με προϊόντα τα οποία, έχουν, τα οποία είναι γενετικά τροποποιημένα. Έχουμε στις 28 Ιουλίου του 2016 αλλά και το 2018 έχουμε την επανέκδοση της άδειας δεν λοιπόν φάνηκε κανένας ε, κίνδυνος ε, σχετικά με την ε, υγεία των ανθρώπων ή για το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, εάν η ΕΦΣΑ θεωρεί ότι ένα γενετικά τροποποιημένο προϊόν είναι ασφαλές, τότε θα πρέπει να πιστεύουμε τα επιστημονικά δεδομένα και γι' αυτό το λόγο δεν θεωρούμε ότι η ε, Επιτροπή ε, ξεπέρασε την δικαιοδοσία της και τις αρμοδιότητες της. Η επιστήμη είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να βασίζουμε τις ε, αποφάσεις μας. Αν λοιπόν δεν ακούμε τη συστάση της ΕΦΣΑ, τότε γιατί την έχουμε. Υπάρχουν επίσης ε, αποφάσεις διακηρύξει, οι οποίε δεν υποστηρίζονται από δεδομένα. Για παράδειγμα ότι αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη χρήση των ε, ε, γλυφοσυνικών. Αυτό όμως το υποστηρίζουν χωρίς να χρησιμοποιούν καθόλου αποδείξεις και επιχειρήματα. Αυτή η αραβόσιτη λοιπόν, αυτά τα είδη αραβοσίτου ε, είναι ανθεκτικά σε συγκεκριμένα παράσιτα και έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε λιγότερα παρασιτοκτόνα και είναι καλό λοιπόν το ότι κάνουμε αυτή τη ε, συζήτηση σήμερα για να μπορέσουμε ε, να συζητήσουμε για αυτό τον σκεπτικισμό που υπάρχει στην επιστήμη. Θα πρέπει να ακούμε τις επιστημονικές αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή, παρακαλώ. Κυρία Ιρλικάρ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μας δίνεται την ε, δυνατότητα να απαντήσουμε σε αυτές τις δύο αντιρρήσεις. Ε, έχουμε δύο είδη ε, γενετικά τροποποιημένου ραβοσίτου. Το ένα αφορά μια άδεια και το άλλο ανανέωση άδεια που χρησιμοποιείται για ζωοτροφές. Θα ήθελα λοιπόν να σας διασφαλίσω ότι όλα τα διαδικαστικά βήματα τα οποία ορίζονται από τους ε, κανονισμούς ε, σχετικά με τα γεννητικά τροποποιημένα έχουν ακολουθηθεί και στις δύο περιπτώσεις. Η ΕΦΣΑ από την πλευρά της έκανε αξιολόγηση αντικτύπου ε, σχετικά με τα πέντε γεγονότα και κατέληξε ε, στην, ε, σε, έδωσε θετική απόφαση σχετικά ε, με τις επιρροές που θα έχει για το περιβάλλον για την ανθρώπινη υγεία. Τώρα όσον αφορά για το είδος για το οποίο υπάρχει αίτηση ανανέωσης ήδη έχει διακηρυχθεί ασφαλές και γι' αυτό και είχε δοθεί άδεια και δεν έχουν ταυτοποιηθεί νέες πληροφορίες οι οποίοι ίσως να άλλαζαν την αρχική αισιόδοξη θετική απόφαση. Όλα τα σχόλια και οι απαντήσεις ε, του ΕΦΣΑ έχουν ε, απαντηθεί και στις ε, δύο περιπτώσεις ακολούθησε δημόσια διαβούλευση και εκεί δεν υπήρξαν κάποια αρνητικά προβλήματα οπότε με βάση τις αποφάσεις τις οποίες ψηφίσαμε 11 Σεπτεμβρίου του 2018 από την αντίστοιχη μόνιμη επιτροπή και αυτό ε, έγινε ε, λόγω ε, πολιτικών αποφάσεων και αρνητικής δημοσιότητας ε, που ακολούθησε αυτό. Οπότε λοιπόν σύμφωνα με τον ε, κανονισμό των επιτροπολογιών και τον κανονισμό για τα γενετικά τροποποιημένα η Κομισιόν, η Επιτροπή θα παρουσιάσει στις 22 Οκτωβρίου το προσχέδιο της απόφασης της στην Επιτροπή. Τώρα υπήρξαν κάποιες ανησυχίες στη συζήτηση που ακούστηκε ε, σχετικά με την ανθεκτικότητα των προϊόντων αυτών θα ήθελα να τονίσω ότι η έγκριση των παρασιτοκτόνων ε, καθώς επίσης ε, και το ανώτατο επίπεδο ασφαλών υπολοιμάτων υπόκεινται στην αντίστοιχη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των φυτών καθώς επίσης ε, και την νομοθεσία σχετικά με τα ανώτατα επίπεδα υπολοιμάτων. Τώρα όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα και τις τρίτες χώρες και τη χρήση παρασυντικοκτώνων εκεί προφανώς η απόφαση να επιτρέψουμε τέτοια καλλιέργεια και την πιθανότητα χρήσης παρασυντικοκτώνων κτόνων επαφίεται σε αυτές τις τρίτες χώρες και δεν μπορεί να νομοθετηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να δώσω έμφαση όμως ότι, στο ότι όσον αφορά το ε, ορισμό επίπεδου ε, υπολοιμάτων θα πρέπει αυτό να ε, σέβεται την υγεία των καταναλωτών θα, η Επιτροπή θα εκδώσει απόφαση ε, μέχρι ότου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η Επιτροπή ε, έκανε μία πρόταση που επιτρέπει τα κράτη-μέλη να περιορίσουν ε, την εισαγωγή γενετικών τροποποιημένων προϊόντων. Κάτι τέτοιο έχει απορριφθεί όμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεχίζουμε λοιπόν να προσδοκούμε τις ε, συζητήσεις ε, μαζί σας όσον αφορά τώρα τις ε, συζητήσεις για την διαφάνεια των δεδομένων και των μελετών που χρησιμοποιήθηκαν. Εκεί θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή έχει κάνει μια φιλόδοξη πρόταση σε αυτό το πλαίσιο για αυξημένη διαφάνεια στο πλαίσιο της αξιολόγησης αντικτύπου που γίνεται από την ΕΦΣΑ και η πρόταση αυτή ε, επεξεργάζεται, την επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και φυσικά η Επιτροπή θα συνεχίσει τις συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Εν κατακλείδη λοιπόν θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν υπάρχει λόγος απόσαρσης αυτών των αποφάσεων καθώς όλες οι διαδικασίες οι οποίες ορίζονται από τον κανονισμό για τα, ε, για τα γεννητικά τροποποιημένα έχουν ακολουθεί και η Επιτροπή ε, σεβάστηκε και στις δύο περιπτώσεις όλες τις διαδικασίες. Επίσης θα ήθελα να ε, επαναλαμβάνω ότι, να επαναλάβω ότι το δικαίωμα ε, εξέτασης από το ε, Κοινοβούλιο αφορά την, την βασική πράξη, το οποίο δεν συνέβη εμπροκειμένο, οπότε παρόλο που η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει εξηγήσεις για τη συγκεκριμένη απόφαση, παρόλο αυτά εμείς ε, οι εξηγήσει που σα δώσαμε ελπίζουμε να βοήθησαν ε, να διασκεδαστούν οι ανησυχίε σα. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους πήραν ε, μέρος στη συζήτηση αυτή. Ας κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα μέχρι τις 10 που θα ξεκινήσει η ψηφοφορία.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

Ja.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

Καλημέρα σε όλους. Αν θέλετε να καθίσετε και να ετοιμάσετε την ε, κάρτα σας για να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία, τις ψηφοφορίες. the first vote Λοιπόν, η Μεταβατική Συμφωνία των Διαθεσμικών Διευθετήσεων για την έδρα του Οργανισμού Φαρμάκων. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ. And it is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. για την αντίρρηση. Για τον κανόνα 106 για τα γενετικό τροποποιημένα αραβοσίτου κτλ. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. And it is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα επίσης επί αντιρρήσεως υπό τον κανόνα 106 επίσης για τα γενετικό στραοποιημένα η δεύτερη αντίρρηση, εν πάση περιπτώσει, άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Θέλατε κάτι να πείτε? Ναι, Πρόεδρε. Δεν λειτουργεί η κάρτα μου. Δεν μπορώ να ψηφίσω. Α, ούτε δίπλα δεν μπορείτε. Μάλιστα. Το Brexit ήρθε νωρί για μένα, Πρόεδρε. Λοιπόν, η Πρόεδρο στο μεταξύ λέει πέρα τη είναι κρίθη. Now we vote on a draft opinion. Σχέδιο έκθεσης για την διάμεση έκθεση του ΠΔΠ 21 Ξεκινούμε με την τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμό 35 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Mrs. Gerling, you are... Η κυρία Γκέρλινγκ. Πέρασε. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Το δεύτερο τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε μου ζητάνε. Καλώς. Άρχεται. And it's closed. Πέρας. Μαζί με την ψήφο της κυρίας Γκέρλιν κατά απορρίπτεται. In, uh, compromise five, we have στη συμβαστική 5 έχουμε προφορική τροπολογία του εισηγητή. Θέλετε να την εισαγάγετε. Ε, απλώς, ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Να μην έχουμε παραπομπή στο EHA και το EA γιατί πιο κάτω ε, αναφερόμαστε στους οργανισμούς, δεν χρειάζεται να το κάνουμε δύο φορές. Μάλιστα, σε ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Έχουμε αντίρρηση για την προφορική. Μάλιστα. Επομένως, μαζί με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά... Κοιτάξτε, χρειαζόμαστε τέσσερις αντιρρήσεις όμως, συνάδελφε. Κάτι λέγεται εκτός μικροφώνου. Για την προφορική Έχετε αντίρρηση. Α, τότε πρέπει να ψηφίσουμε χωρίς την προφορική τροπολογία. Ε, κύριε Πιέκα, μόνο εσείς σηκώσατε το χέρι σας και εγώ θεώρησα ότι υπάρχει μία αντίρρηση και μόνο. Θέλετε κάτι να πείτε. Ζητώ συγγνώμη, ε, πρόεδρε, στα πολωνικά θα μιλήσω. Κοιτάξτε, όταν έχουμε συμβιβαστική τροπολογία, η προφορική κατά τη διάρκεια της ψήφου δεν είναι σωστή. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει την ώρα που συζητεί το ο συμβιβασμός. Με συμβιβαστική δεν μπορεί να γίνει περαιτέρω διόρθωση. Δεν είναι αποδεκτό αυτό. Θέλει να απαντήσει ο ηγητής. Ναι, πρόεδρε, δεν πρόκειται για πρόταση του εισηγητή εδώ άλλης ομάδας του Κοινοβουλίου που ε, λάβαμε υπόψη την άποψή τους και δεν πρόκειται για ουσιαστικό θέμα. Και μάλιστα γλωσσικό είναι. Έχουμε παραπομπή σε όλους τους οργανισμούς τους απαριθμεί ο εισηγητής, είναι στη συμβαστική και δύο εξ αυτών μόνο σε αυτό το δεύτερο σημείο, σημείο ε, ε, αναφέρονται δεύτερη φορά. Αν δείτε τη συμβαστική όμως ε, τροπολογία, καλύπτονται όλοι οι οργανισμοί. Αναφερόμαστε σε όλους αυτούς. Το είχαμε συζητήσει και με άλλες ομάδες. Και είναι πραγματικά συντακτικό, γλωσσικό θέμα δηλαδή. Δεν ήταν καν δική μου πρόταση, απλώς την έλαβα υπόψη μου εχθέ γιατί ήταν σωστή. Δεν αποσύρουν την αντίρρησή τους οι συνάδελφοι παρόλα αυτά, λέει ο Πρόεδρος. Τη διατηρούν διατηρούν την αντίρρησή τους. πόσοι, έχουν αντίρρηση στην προφορική τροπολογία, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι τους. Μάλιστα. Καλώ. Άρα συμβαστική χωρί την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται.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 αποχές εγκρίνεται. Επομένως ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την γνωμοδότηση άρχεται ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα για το σχέδιο έκθεσης όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Ξεκινάμε με την τροπολογία 24 παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμ... Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρτη ψηφοφορία. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Συμβαστική τροπολογία είναι να συνελέγξουμε καλύτερα. Άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Και εγκρίνεται. Περνάμε στην ε, σελίδα 4. Τροπολογία 181 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3α τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε σε 7. Συμβαστική 2α. Υπέρ παρακαλώ. Συμβαστική 2α. Υπέρ παρακαλώ. Συμβαστική 2α. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29 τώρα, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 29. Νομίζω ότι απορρίπτεται, λέει η Πρόεδρος. Αλλά νωρίτερα έκανα λάθος εκτιμήσεις μου. Πέρας. Και γκρινεται 193 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2β υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε σε λίδα 11 τώρα. 2.29 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 226 και τραν 28 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ...2, 22, 23 και 3.27 μαζί υπέρ παρακαλώ. Στη σελίδα 12 είμαστε λέει πρόεδρος. Απορρίφθηκε η συμβαστική τροπολογία, επομένω θα πρέπει να ψηφίσουμε τώρα κάθε επιμέρου τροπολογία ξεχωριστά. Ξεκινάμε με τη 222, 223 και την τράν 27 από κοινού υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ απορρίπτονται. Τροπολογία 227, 365, 373 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτονται. 228, 230, 368 και 370 μαζί υπέρ παρακαλώ κατά. Αποχές απορρίπτονται. 369, 371, 372 υπέρ παρακαλώ κατά. Αποχές απορρίπτονται. Αλεκτρονικός έλεγχος. Άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. And it's closed. Πέρας. Απορρίπτονται. 219 καταπίπτει. 218 και τραν 26 μαζί υπέρ παρακαλώ κατά. Αποχές απορρίπτονται. 217 υπέρ παρακαλώ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τραν 29 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πάμε σελίδα 17 λέει πρόεδρος. 36 υπέρ. Ψηφίζουμε τροπολογία 36 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία. Διακόπτη προέδρο. Οι σοσιαλιστές ήταν υπέρ ή κατά. Το EPP, το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστέ είναι κατά. Θέλετε παρόλα αυτά να ελέγξουμε την τροπολογία 36. Ας την ελέγξουμε, ας την ελέγξουμε άμα θέλετε. Άρτη ψηφοφορία. Ελεκτρονικό έλεγχο για τροπολογία 36, άρχεται Πέρα. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4α, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. Πάμε σελίδα 19. Συμβαστική 4β υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. Συμβαστική 4c υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 358 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 302 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 312 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 314 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ΕΛΚ πως ψηφίζει υπέρ ηλεκτρονική επαλήθευση ήταν, δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 315 υπέρ. Κατά. Αποχές Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 315, άρτη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 316 πέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για 316, άρτη ψηφοφορία. Μάλλον το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε με την προηγούμενη πέρας και όντως απορρίπτεται. 8α συμβαστική υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8β συμβαστική. Α, μα καταπίπτει, διορθώνει πρόεδρος. Συμβαστική 9 στη σελίδα 26 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει και ψηφίζουμε έτσι την τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε τις ακόλουθες. 356 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 361 και 362 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 363 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 364 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 366 και 367 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 374 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Πάμε σελίδα 32 391 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 392 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 τώρα. 74 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 74 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. και γκρίνεται. 75 τώρα υπέρ κατά οι σοσιαλιστές πως ψηφίζουν υπέρ μάλιστα γκρίνεται. τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση τροπολογία 2 άρχιτη ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τραν 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4. Την 76 ψηφίσαμε, λέει πρόεδρος. Με εγκρίναμε την τραν 1. Σα το συγγνώμη. Ψηφίζουμε μόνο το πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την 76. Οι σοσιαλιστές ήταν κατά, τέλος πάντων, πέρας ψηφοφορίες και όντως απορρίπτεται. Τροπολογία 4 τώρα, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 και τραν 2 μαζί υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνονται 6 υπέρ. Κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 6. Πέρας και εγκρίνεται. 78-79 μαζί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Τραν 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 80 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν ψηφίσαμε την τραν 4, σας το συγγνώμη, λέει πρόεδρος. Τραν 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Τραν 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 και 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 101 και τροπολογία 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τραν 13 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται τραν 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τραν 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 και 108 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία άρθρη ψηφοφορία παρακαλώ πέρας και εγκρίνεται Okay, so this concludes the voting uh, session. Mr. Is coming. And uh, next item is the... Λοιπόν, έχουμε τώρα την ακροματική διαδικασία του Bernard Ουλ, διοικητικού διευθυντή της ΕΦΣΑ για προκειμένου να ανανεωθεί η εντολή του, ίσως σε 15 λεπτά. Α, όχι, είναι ήδη εδώ. Σε 5 λεπτά Uh, Σε πέντε λεπτά θα είναι εδώ. Παρακαλώ μείνετε στην αίθουσα.

Okay. Let's start the, the meeting. Να συνεχίσουμε. Θα ακούσουμε τον κύριο Μπερνάρντ Ουλ, διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΦΣΑ. Το, συμβου, το Συμβούλιο της ΕΦΣΑ αποφάσισε να παρατείνει τη θητεία του σε συνάντηση 10 Οκτωβρίου. Τον Ιούνιο του 2014 ανέλαβε τα καθήκοντά του ο κύριος Ουλ, εκτελώντας χρέη του συμβούλου τους τελευταίους μήνες. Καθότι τον γνωρίζουμε, τον κύριο Ουλ, ε, χρησιμοποίησαμε μια απλουστευμένη διαδικασία και όχι επίσημη, αν θέλετε, ακροαματική διαδικασία. Μια απλή ανταλλαγή απόψεων Επομένως η σημερινή παρουσία, συνάντηση, είναι απλώς μια ανταλλαγή απόψε με τον οργανισμό. Μπορούμε να συζητήσουμε το πρόγραμμα και τους στρατηγικούς του στόχους, του οργανισμού δηλαδή, μέχρι το 2020 και χωρίς άλλη καθυστέρηση τώρα, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ουλ των οποίων καλωσορίζω. Και θα παρακαλούσα οι συνάδελφοι να μας γνωστοποιήσουν αν θέλουν να μιλήσουν. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα και ο πλευρά μου, αξιότιμα μέλη, ε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την δυνατότητα σήμερα να σας κάνω μια δήλωση και να ακούσω τις ερωτήσεις σας αν έχετε. Με τιμά το να είμαι υποψήφιος ε, για ανανέωση της ε, θητείας μου ως ε, διευθύνων σύμβουλος του ΕΦΣΑ. Ε, ξέρω ότι το ξέρετε, αλλά ας επαναλάβουμε τη βασική αποστολή του ΕΦΣΑ. Είναι η παροχή των καλύτερων δυνατών επιστημονικών συμβουλών για την, κυρίως για την ασφάλεια τροφίμων, για την υγεία των ζώων και των φυτών και για αναδυόμενους κινδύνους αυτός είναι ο βασικός στόχος, η βασική αποστολή μας. Και πώς παρέχουμε αυτή την προσθέμενη αξία για τους ηθήνοντες της πολιτικής και τους πολίτες, παρέχουμε επιστημονικές συμβουλές για τους κινδύνους, χημικούς, βιολογικούς, για την ευζοία των ζώων, για την υγεία των φυτών, εκτιμήσεις ασφαλείας για τα τρόφιμα πριν την απελευθέρωσή τους, ετήσιες εκθέσεις που επίσης είναι σημαντικό μέρος της δουλειά μας ε, για κατάλοιπα για την μικροβιακή αντοχή Αυτά αποκινούμε άλλους οργανισμούς με το Κέντρο Ελέγχου των Νόσων στο Χόλμη και με τον Οργανισμό Φαρμάκων στο Λονδίνο. Επίσης φιλτράρουμε αν θέλετε ενδεχόμενους αναδυόμενους κινδύνους στην αλυσίδα τροφίμων ώστε να τους εντοπίσουμε και να τους αντιμετωπίσουμε πριν την εμφάνισή τους και ενημερώνουμε με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο και τους καταναλωτές και τους υπευθύνους, τους αρμοδίους. Πριν από κάποια χρόνια, ήταν τον Απρίλιο του 2014, ε, στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΝΒΗ, της εντολής πριν από τη δική σας στο Στρασβούργο που είχα την τελευταία μου ακροαματική διαδικασία ως ε, νεοεκλεγής διευθύνων σύμβουλος και είχα επιλέξει τέσσερις θεματικές σωστές επιστημονικές συμβουλές ανάπτυξη του θεματολογίου της ε, ανάλυσης κινδύνου οικοδόμηση διαφάνειας και επικοινωνία. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να εκτιμήσω κατά πόσον ο ΕΦΣΑ κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτούς τους στόχους. Για το πρώτο, για τα επιστημονικά. Τα πήγαμε καλά με τις επιστημονικές συμβουλές. Αυτά τα 4,5 χρόνια εκδώσαμε πάνω από 2.000 επιστημονικές συμβουλές και το 99,9% θεωρώ δεν είχε κανένα αμφίσιμο ή αντιφατικό θέμα. οι υπεύθυνοι τη αξιολόγηση κινδύνου εφαρμόζουν τις συμβουλές αυτές. Έχουμε μακροχρόνια προγράμματα για πρόσθετα τροφίμων, ε, ε, λιπάσματα, ζυζανιοκτώνα κτλ. Έχουμε εκτιμήσεις ε, ταχείας ε, εκδήλωσης νόσων για τον έμπολα μεταξύ άλλων για παράδειγμα. Ετήσιες επίσης νόσους ε, τον ε, αφρικανικό ε, πυρετό των χείρων για παράδειγμα ξυλέλα φαστιντιόζα τις ε, ασθένειες των, της ελιάς υπό το νέο καθεστώς δηλαδή της υγείας των φυτών και στο πλαίσιο ίσως όχι σε τόσο θέση προσκυνείου εξεργαζόμαστε και έγγραφα καθοδήγησης που είναι τα εργαλεία της αξιολόγησης του κινδυνού που εξηγούν δηλαδή πώς προχωρούμε σε αυτή την αξιολόγηση. Έχουμε μεγάλη δέσμη τέτοιων εγγράφων, θα αναφέρω απλώ τρία. Είναι η αβεβαιότητα στην αξιολόγηση κινδύνου. Πώ χειριζόμαστε την αβεβαιότητα επιστημονικά. Ήταν τεράστιο έργο τη Επιτροπή μα Επιστημονική τελευταία χρόνια. Είμαστε πάντα βασισμένοι στι επιστημονικέ ενδείξει με μελέτες που μας δίνει ο κλάδος αλλά και ακαδημαϊκές πηγές και βεβαίως βιολογική σχετικότητα των αντικτύπων, χρησιμότητα. Τώρα, οι επιστημονικές μας συμβουλές είναι επικαιροποιημένε. Εκτός Ευρώπης, όταν συναντούμε τους ε, συνομολόγους μας από την Κίνα, από την Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, Έχουμε πολύ θετικά σχόλια για την επιστημονική ποιότητα της δουλειάς μας. Και κάποιες χώρες σχεδόν ανοιχτά μας λένε, εμείς δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά, απλώς παίρνουμε τη δουλειά της, του ΕΦΣΑ ως πρότυπο για να προχωρήσουμε. Επομένως αυτό είναι, αυτό είναι καλό σημάδι ότι η επιστήμη που χρησιμοποιεί ο ΕΦΣΑ είναι επικαιροποιημένη και χρησιμοποιείται ως πρότυπο. Για να επανέλθω λοιπόν στο Κοινοβούλιο, νομίζω ήταν πολύ σοφή από, απόφαση του 2002 όταν υιοθετήθηκε ο γενικό ε, κανονισμός για τα τρόφιμα να δημιουργηθεί ένας ε, μικρό οργανισμός με 450-500 ανθρώπους προσωπικό. Αυτό το πρότυπο των κρατών μελών που έχουν τις εμπειρογνώμονες και που μας τους παρέχουν εθελοντικά πάνω κάτω είναι ένας ευέλικτος και ευφυής τρόπος και όχι ιδιαίτερα επαχθής τελείω διαφορετικό από το αντίστοιχο πρότυπο των Αμερικανών και κοιτώντα πίσω 15 χρόνια είναι απίστευτο με 18 μόλι εκατομμύρια ευρώ το έτος τι καταφέραμε. Αν δείτε την FDA την Αμερικανική ή την e DPA το περιπολογισμό του είναι μεταξύ 5 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων με άνω των 10.000 υπαλλήλου. Είμαστε ένα μικρό οργανισμό και μπορούμε και κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε μόνο και μόνο λόγω του ενθουσιασμού των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών. Και για μένα είναι μεγάλη ικανοποίηση που βλέπω τον ενθουσιασμό των συναδέλφων αυτών για τα της ασφάλειας των τροφίμων και για την εθελοντική συνεισφορά των κρατών μελών βεβαίως είμαι ευγνώμων και αυτό είναι πραγματικά ένα παράδειγμα της Ευρώπης εν δράση. Ένα από αυτά που έλεγε ο Ρομπέρτ Σουμάν. Δηλαδή ένα απτό παράδειγμα ευρωπαϊκής κοινή δράσης και ολοκλήρωσης. Τώρα το δεύτερο που ανέφερα πριν, κατά πόσον υλοποιήσαμε το θεματολόγιο αξιολόγηση κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κάναμε αυτό με συμβουλευτικό φόρουμ, με τα σημεία επαφή που είχαμε στα κράτη-μέλη και τώρα Εργαζόμαστε επί κοινών έργων για ιούς, για τον καμπυλομπάκτερ μέχρι ε, ασκήσεις ε, ετοιμότητος ε, κινδύνου. Και ευχαριστώ όλους τους εταίρους και τα κράτη-μέλη για την συνεχιζόμενη στήριξή τους στον ΕΦΣΑ. Για το τρίτο σημείο για τη διαφάνεια, την ε, ανεξαρτησία. Ξεκινήσαμε αυτόν τον αγώνα το 2014 για έναν ανοιχτό και ανεξάρτητο ΕΦΣΑ, ώστε να έχουμε τις μεθόδους και τα δεδομένα μας δημοσίως διαθέσιμα για να μπορεί να τα ελέγχει οποιοδήποτε και να αντιγράφει τις επιστημονικές συμβουλές μας. Υλοποιήσαμε άνω των 35 μέτρα, υλοποιήσαμε νέα πολιτική ανεξαρτησίας, εξασφάλισης ανεξαρτησίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την ε, ε, συμβουλή της που συνοδεύεται και από επικρίσεις επικοδομητικές σε σχέση με θέματα δημοσιονομικά προϋπολογισμού, δηλαδή συναλλαγές. Είχαμε τα τελευταία πέντε έτη πράσινο φως, θετικό δηλαδή πόρισμα και από την Επιτροπή Προϋπολογισμού Εφαρμόσαμε επίσης μια προσέγγιση για τους ενδιαφερόμενους φορείς με άνω των 100 φορείς που είναι εγγεγραμμένοι πλέον στο δίκτυό μας και προχωρούμε για να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη διάδραση με την κοινωνία των πολιτών. Αυτό μας ε, επέτρεψε μια μοναδική πρωτοβουλία μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι η εταιρική σχέση για την υγεία των μελισσών για να συλλέγουμε δεδομένα ώστε να κατανοούμε καλύτερα τις πιέσεις που ασκούνται στα μελίσια στις μέλισσες. Και πολύ μας ικανοποιεί ότι λάβαμε εντολή από το Κοινοβούλιο να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι απόδειξη εμπιστοσύνης για τη δουλειά μας. Επίσης ε, για την... ένα άλλο έργο στην, υγεία, στην ευζοία των ζώων ήταν για τα κουνέλια των καλλιεργιών. Υπό την έννοια της διαφάνειας και του ανοιχτού μας χαρακτήρα είναι περισσότερο προϋπόθεση για την υπευθυνότητα, για την ευθύνη που πρέπει να έχουμε, γιατί βεβαίως είμαστε υπεύθυνοι έναντι των κρατών μελών και θεσμικών οργάνων για τον προπολογισμό που λαμβάνουμε από τους φορολογουμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ανακοίνωση στα θέματα επικοινωνίας ε, ήταν από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε. Με τόσους πολλού φορεί διεθνώ και τόσα πολλά μέσα. Εμείς έχουμε ένα, μια ορθολογική προσέγγιση με ομάδες στόχου καλά αναλυμένες αν θέλετε στοχευμένες και καλή συνεργασία με τις αρχές ε, διαχείρισης του κινδύνου. Με όλα αυτά μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι θα έλεγα και ναι και όχι. Ναι, διότι το έργο του ΕΦΣΑ έχει συνεισφέρει σημαντικά στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε παγκόσμιος πρωταθλητής στα αγροτρόφιμα έχουμε συνεισφέρει σε ένα υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητος αυτό το έδειξε και η άσκηση Refit του 1978, με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων φορέων, αλλά δεν μπορούμε να είστε ικανοποιημένοι. Έχουμε ακόμα πολλές νόσους, έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τη μικροαιακή αντοχή, έχουμε διάφορες νόσους φυτών και ζώων που πλήττουν. Πιο συγκεκριμένα δεν υπήρξαμε πάντοτε επιτυχής στην επικοινωνία των επιστημονικών μας ενδείξεων και η μέθοδοι μας δεν μας επέτρεψε να είμαστε τόσο ανοιχτοί όσο θα επιθυμούσαμε. Και εδώ θα σχολιάσω μια πρόσφατη εξέλιξη. Είναι και ο λόγος για τον οποίο ήμασταν τόσο θετικοί με την πρόταση διαφάνειας και βιωσιμότητας. Θα είχαμε τη νομική βάση και τους πόρους για να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα προς μεγαλύτερη διαφάνεια. Και όσο νωρίτερο εγκριθεί η πρόταση αυτή τη Κομισιόν από του νομοθέτε, τόσο το καλύτερο για τη δουλειά μα. Δημιουργήθηκαν προσδοκίε από την Επιτροπή BEST για καλύτερη προσβασιμότητα στα δεδομένα. Κατανοούμε βεβαίω ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία απαιτεί χρόνο για ποιοτικά αποτελέσματα. Το κατανοούμε, το αναγνωρίζουμε. Δεν είμαστε οι νομοθέτες. Είμαστε απλώς το μέσον. Παρόλα αυτά θα σας ζητούσα στο φάκελο αυτό να δώσετε την υψηλότερη δυνατή προτεραιότητα όχι μόνο για το καλό του ΕΦΣΑ αλλά για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών για καλύτερη διαφάνεια και καλύτερη αξιολόγηση κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων. Σας ευχαριστώ για τη συνεχιζόμενη δέσμευση στο φάκελο αυτό και για έγκαιρη συμφωνία. Έχω ακόμα δύο λεπτά, Πρόεδρε. Ωραία. Οι μεγαλύτερε προκλήσει για τα επόμενα χρόνια θα είναι οι πόροι, η χρηματοδοτική και οι πόροι οι ανθρώπινοι ως προς την εμπειρογνωμοσύνη γιατί ο ΕΦΣΑ δεν θα μπορέσει με αυτό τον προϋπολογισμό να μπορεί να παραδίδει και στο μέλλον. Έχουμε ακόμα πρικλέσεις ε, στα επίπεδα της χημίας ε, και της ε, συνθετικής ε, βιοχημίας. Η επικοινωνία όλων αυτών των επιστημονικών ενδείξεων εξακολουθεί να είναι πρόβλημα, πρόκληση και η ετοιμότητα, η προετοιμασία για τις άγνωστες τάσεις του μέλλοντος. Θα χρειαστούν διάφορες πρωτοβουλίες που θα τις καταδείξουμε στη στρατηγική 2027 του ΕΦΣΑ όπως τον ονομάζουμε αλλά αυτό που συνδέει την αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων είναι αυτό που εμείς νομίζουμε απεριόριστη συνεργασία. Και χρειάζεται σε όλα τα επίπεδα εντός της του ΕΦΣΑ με τους συναρμόδιους των κρατών μελών, με νέους οργανισμούς που υποβάλλουν στοιχεία στην Επιτροπή ΕΝΒΗ αυτοί, οι 45 οργανισμοί και υπηρεσίες δεν θα μπορούσαν να οικοδομήσουν έναν οργανισμό One Health, όπως θα τον έλεγε κανείς. Ίσως να ήταν μια ιδέα. Αυτό ισχύει και για την Γαμαδέλτα Σάντε, την Άγκρη, την Connect, τις Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής δηλαδή, και πρέπει και να συνεργαζόμαστε και με το Κοινοβούλιο, γιατί είμαστε εδώ να σας παρέχουμε συμβουλές και βεβαίως με τους ε, διεθνείς εταίρους μας. Χρειαζόμαστε παγκόσμιες προσεγγίσεις στην αξιολόγηση του κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. Και βεβαίως πρέπει να ενσωματώσουμε τις κοινωνικές επιστήμες περισσότερο στη δουλειά μας για να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογική καινοτομία, το crowdsourcing, το cloud computing κτλ. Για τους πόρους θα ζητήσουμε την υποστήριξή σας για μεγαλύτερο προϋπολογισμό στο μέλλον για τον ΕΦΣΑ. Επαναλαμβάνομαι ίσως, αλλά φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τις, τις προσδοκίες των πολιτών με τον προϋπολογισμό των 80 εκατομμυρίων που έχουμε. Ήταν τιμή πάντως και προνόμιο για μας που συνεργαστήκαμε μαζί μας. Μερικές φορές είχαμε δύσκολες συζητήσεις και παθιασμένες αλλά ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις είχα πάντοτε την αίσθηση μιας ενότητος για τον συνολικό στόχο που είναι η ασφάλεια των τροφίμων για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι μεγάλη χαρά να, συνεχίσουμε, να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί σας τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, δόκτωρα Ε, Και τώρα ε, η κυρία Γιούσο Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος της κυρίας Αγιούζο, η οποία δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα. Κύριε Ούρλα, καταρχάς σας καλωσορίζω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και σας συγχαίρω ειλικρινά για την για τον διορισμό σας που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΣΑ σε σχέση με την ανανέωση της θητείας σας. Σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες που έχετε βάλει προκειμένου να γίνει γνωστή η συμβολή θετική της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων και γιατί μας δίνετε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε πώς λειτουργεί καλύτερα ο οργανισμός αυτός. Ως εκτελεστικός διευθυντής έχετε κάνει μια ήδη σημαντική εργασία και καταφέρατε να διαχειριστείτε καταστάσεις δύσκολες. Είμαι πεπισμένη ότι θα συνεχίσετε να καταβάλλετε προσπάθειες για τη βελτίωση της αρχής αυτής και κατά τη διάρκεια της επόμενης θητείας σας εφόσον αναθεωθεί. Μία απλή ερώτηση θα ήθελα να θέσω ολοκληρώνοντας, αλλά πολύ σημαντική. Ε, γιατί έχει να κάνει με τις πολλές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε. Εφόσον ανανεωθεί η θητεία σας για πέντε ακόμα χρόνια, ποια θα είναι η βασική σας προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρο. Και, εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στα μέλη. Ορισμένοι ήδη ε, ζήτησαν το λόγο. Κύριε Πόρτς. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Πιστεύω ότι αναμφίβολα είστε το κατάλληλο άτομο να γεννηθείτε της υπηρεσίας και αποδείξατε επανειλημμένως στην ε, δέσμευσή σας ε, για την δουλειά. Έχετε καλές επικοινωνιακές ικανότητες ε, και πιστεύω ότι είστε πολύ καλός για τη συγκεκριμένη θέση, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι ικανοποιημένο με όλα όσα έχουν γίνει. θα περίμενα να είχατε πει όχι μονάχα για τις επιτυχίες αλλά και για τα λάθη διότι όλοι κάνουν λάθη και εσείς δεν αναφέρατε ούτε ένα και για μένα λοιπόν θα ήταν ενδιαφέρον το τι πιστεύετε για τα λάθη που έχουν γίνει όχι από εσάς προσωπικά αλλά από την υπηρεσία σας γενικά για παράδειγμα η αξιολόγηση των κλειβαστικών, ε, των γλυκαντικών, πώς θα το κρίνατε αυτό. Η Επιτροπή σας πείσε να κάνετε μη επαναξιολόγηση. Είναι περίεργο όλο αυτό λοιπόν. Το επόμενο σημαντικό ερώτημα για μένα είναι η διπλή πορεία όσον αφορά την αξιολόγηση και την, αξιο... την αδειοδότηση ορισμένων ουσιών. Ίσως καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι αξιολογεί τα ζυζανιοκτώνα, τα παρασυντοκτώνα μία υπηρεσία και άλλες ουσίες μία άλλη υπηρεσία. Είναι περίεργο λοιπόν αυτή η διπλή διαδικασία, αυτή η επικάλυψη. Και ορισμένες φορές είναι πολύπλοκο, όχι μόνο για μας, αλλά και για το ευρωπαϊκό κοινό και τις υπηρεσίες. Επίσης όσον αφορά την ε, πρόταση για τα γενετικά τροποποιημένα και νομίζω ότι η εισηγήτρια θα αναφερθεί σε αυτό. Έχουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, δύο εναλλακτικέ. Μία φορά είτε τα αγροκτήματα, είτε να το κάνουμε γρήγορα, είτε να το κάνουμε καλά. Λοιπόν, ε, σε οτιδήποτε, είτε θα το κάνεις καλά, είτε θα το κάνεις γρήγορα. Ε, και τι προτιμάτε λοιπόν, να γίνεται γρήγορα ή να γίνεται καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάισνα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ κύριε για την παρουσίασή σας. Πριν από μερικά ε, χρόνια με την ε, κυρία Γιούσο επισκεφθήκαμε την ΕΦΣΑ και ε, είχα πιστεί με τα όσα είχα δει και οι επιστήμονες με τους οποίους συζήτησα ε, μου είχαν κάνει πολύ θετική εντύπωση. Οπότε προσωπικά θα έλεγα ότι, είναι, ότι είμαι μια φαν του ΕΦΣΑ, όμως ε, ε, είμαι ικανοποιημένη που υπάρχει ο συγκεκριμένος οργανισμός. Είπατε ότι ε, στην επικοινωνία δεν έχετε κάνει αρκετά όσον αφορά την αντιμικροβιακή αντίσταση. Τι θα μπορούσατε να είχατε κάνει. Ε, δεν εισακουστήκατε, δεν ε, ε, δώσατε αρκετές συμβουλές όταν λέτε ότι η επικοινωνία δεν ήταν καλή. Δεύτερον, είπατε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα διαφάνεια, περισσότερα δεδομένα, Οπότε εσείς για να μπορείτε να δώσετε περισσότερα δεδομένα χρειάζεστε περισσότερα χρήματα. Τι χρειάζεστε για να το κάνετε αυτό. Και επίσης είπατε ότι τα 80 εκατομμύρια δεν είναι αρκετά, το καταλάβαμε αυτό. Πόσα Λοιπόν, ε, χρειάζεστε, δεν παζάρει εδώ πέρα, όμως ε, τι ε, περισσότερα θα μπορούσατε να κάνετε εάν είχατε περισσότερα χρήματα, πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε περισσότερο τους, Ευρω... τους Ευρωπαίους πολίτες, τι θα άλλαζε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Άουσλινγκ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και για τη δήλωσή σας. Κατανοούμε ότι ε, η ΕΦΣΑ είναι ένας σημαντικός οργανισμός που θέλουμε να ενισχύσουμε και συνεισφέρατε σε αυτό. Βέβαια έχετε μία ε, ουδέτερη στάση και έτσι πρέπει άμα καθώς ήσασταν από αυτήν την πλευρά των εδράνων θα μπορούσατε να το κάνετε αυτό. Όμως είχατε κάνει κάποιες ε, δηλώσεις που, ήταν, ε, που προκάλεσαν αντιδράσεις όπως ε, για παράδειγμα το, η απόφαση για το γλυφοσάτ ήταν λοιπόν όλα αυτά πράγματα στα οποία μπορούμε να είμαστε επικριτικοί και δώσατε μια συνέντευξη σε, αυστριακή, σε ένα αυστριακό περιοδικό και είπατε ότι η παραδοσιακή γεωργία δεν είναι αποτελεσματική και ότι χρειαζόμαστε πιο εντατική ε, γεωργία ε, και στην ίδια συνέντευξη είπατε ότι τα γενετικά τροποποιημένα είναι ο καλός δρόμος, οπότε θα πρέπει να τα παρουσιάσουμε καλύτερα. Ήταν μια δήλωση λοιπόν που θα μπορούσαμε να την αντιγράψουμε από μια δήλωση της βιομηχανίας. Οπότε είστε ουδέτερος το βλέπετε, ε, καλό, το βλέπετε καλό όταν για αποφάσει που έχουν προκαλέσει τόσες ε, αντιδράσεις να κάνετε τέτοιε δηλώσεις οι οποίες ε, προκαλούν, αμφισβητούν την εμπιστοσύνη που υπάρχει. Δεν... Μελλοντικά λοιπόν είναι κάτι το οποίο μια στάση την οποία θα αλλάζατε θα ήταν κάπως διαφορετική. Υπάρχει λοιπόν από μερικού έλλειψη εμπιστοσύνη επειδή κάνετε κάποιε πολιτικέ δηλώσει, όπω για παράδειγμα η δήλωση για τα γενετικά τροποποιημένα. Θα πρέπει λοιπόν με κάτι τέτοιε δηλώσει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Οπότε, πώ ορίζετε το ρόλο σα ε, για το μέλλον, θα ε, κάνετε και πολιτικά επιχειρήματα ή θα προτιμάτε να είστε πιο ουδέτερος. Είπατε ξεκάθαρα το τι χρειάζεται μελλοντικά η ΕΦΣΑ, όμω θα ήθελα να αναφερθώ στην οδηγία για την ε, διαφάνεια. Ως ε, πράσινη λοιπόν, θέλουμε να προωθηθεί κάτι τέτοιο. Είχαμε μια συνάντηση χθε για αυτό, όμως υπάρχει πρόβλημα και συμφωνούμε σε αυτό. Όταν η Επιτροπή παίρνει ε, σύντομα αποφάσει. Εμεί έχουμε τρομερή πίεση να εφαρμόσουμε κάτι θα χαιρέτιζα λοιπόν εάν επιτευχθεί στόχος πριν από τις εκλογές, όμως συνολικά πιστεύω ότι ότι και αυτό είναι σημαντικό πέρα από τα χρήματα το ζήτημα της διαφάνειας, ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, ούτως ώστε και οι πολίτες ε, να έχουν εμπιστοσύνη για την υπηρεσία σας. Και τέλος, αυτό το οποίο πρόσεξα τα τελευταία χρόνια είναι ότι σε πολλές αποφάσεις δεν αποκλίνουμε από την αρχή της ε, πρόληψης ε, προς ε, την πρόληψη κινδύνων και αυτό με ανησυχεί σε πολλές αποφάσεις της ΕΦΣΑ. Τι έχετε να πει σε αυτό, ότι ε, το ζήτημα της πρόληψης ε, είναι, δεν πρόκειται να το διαπραγματευτούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μιλιόγα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε κύριε Ουρ, Σας ευχαριστώ όχι μονάχα που ήρθατε, αλλά και για την ε, παρουσίασή σας που αναφερθήκατε σε όλα τα θέματα ε, τα οποία είχατε δηλώσει και στο παρελθόν. Πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι πολύ τυχερή που υπάρχει η ΕΦΣΑ, ότι υπάρχει ένα πολύ ψηλό επίπεδο ασφάλειας τροφίμων στην Ευρώπη και εγώ θα χαιρόμουν αν υπήρχε ανανέωση της θητείας σας και είναι καλό για μια ευρωπαϊκή υπηρεσία όταν υπάρχει ένας ε, χαρισματικός άνθρωπος ε, στην κορυφή της, για να το θέσω έτσι διπλωματικά αναφερθήκατε σε ένα θέμα το οποίο επίσης με απασχολεί αρκετές φορές που είναι οι εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη ε, που, είναι, που βρίσκονται στο... αυτό είναι ο πυρήνας της ΕΦΣΑ ε, συνεισφέρουν σε εκθέσεις ε, που παρουσιάζεται και οι εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη είναι ταυτόχρονα και πρόβλημα. Μιλήσαμε γι' αυτό αρκετές φορές και μεταξύ μας ε, και θα χαιρόμουν ιδιαιτέρως αν ε, θα μπορούσατε να παρουσιάσετε κάποιες ιδέες σχετικά με το πώς μπορούμε να το επιτύχουμε ούτω ώστε οι εμπειρογνώμονες να συνεισφέρουν, να έχουν όρεξη, τα κράτη-μέλη να είναι έτοιμα να επενδύσουν, να δώσουν κάποια χρήματα ή τουλάχιστον να δημιουργήσουν τις δυνατότητες ούτω ώστε οι ειδικοί μερικές φορές να συνεισφέρουν, να έχουν το χρόνο να προετοιμάσουν ε, διότι ε, και ο Μάρτιν μόλις το είπε, το ζήτημα της διαφάνειας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το πόσο ε, ανεξάρτητα και διαφανώς εργάζεται η ε, ΕΦΣΑ. Θα χαιρόμουν λοιπόν αν θα μπορούσατε να αναφερθείτε και σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λίζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ουόλ για την παρουσίαση, για τη δουλειά σας και θα χαιρόμουν αν συνεχίζατε. Όμως θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα. Έχουμε ε, την επανεξιολόγηση του ε, General Food Law Έχουμε τη συζήτηση όσον αφορά το διάγραμμα και πιστεύω ότι θα πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Επιτροπή. Ο τρόπος που δουλεύει η Κομισιόν, η Επιτροπή δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και χρόνια συζητά εσωτερικά αλλά και με τα ενδιαφερόμενα μέρη ε, και όταν ε, κατατίθεται η πρόταση, εμείς μέσα σε τρεις ε, εβδομάδες θα πρέπει να το εγκρίνουμε και κατά προτίμηση χωρίς καθόλου αλλαγές το καλοκαίρι μου είπαν ότι ε, η Επιτροπή δεν χρειάζεται να συζητάμε τα ενδιαφερόμενα. Ότι εμεί δεν χρειάζεται να συζητήσουμε με τα ενδιαφερόμενα μέρη γιατί το έκανε ήδη η Επιτροπή. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Όταν υπάρχει μία πρόταση που θα πρέπει να εγκριθεί πριν από τι εκλογέ, θα πρέπει να παρουσιάζεται και εγκαίρω. Ε, και αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία διάταξη, όταν βλέπουμε το τι έχουμε την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, έχουμε 7-8 αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Θα πρέπει να εξετάσουμε κάθε, ε, κάθε σημείο και έτσι λοιπόν πιστεύω ότι όσον αφορά τον κανονισμό General Food Law θα πρέπει ε, να πάμε αργά και προσεκτικά. Ε, όμως εμείς θα πρέπει ε, να ε, δείξουμε ξεκάθαρα στην Επιτροπή ότι χρειαζόμαστε χρόνο και αν θέλουμε να εγκριθεί κάτι θα πρέπει να το καταθέτουμε και εγκαίρως. Ε, πολλές φορές ε, υπήρχαν ε, θέματα στο σιρτάρι στην Επιτροπή και τώρα ξαφνικά τα θυμάται και πρέπει πριν τον Μάιο, Ιούνιο να τα έχουμε όλα ψηφίσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μελά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Ούρλα που ήρθατε εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξ ονόματος πολιτικής ομάδας. Πολλές ερωτήσεις θα ήθελα να σας θέσω. Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα και ιδίω η σημασία που δίδεται για τη διατροφική ασφάλεια, εσείς πώς εκτιμάτε ορισμένα σημαντικά σημεία της μεταρρυθμίσης αυτής, δηλαδή τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων, το ζήτημα της διαφάνειας, καθώς επίσης και το ζήτημα της διακυβέρνησης, που θα επέτρεπε ενδεχομένω τα κράτη-μέλη να είναι πιο παρόντα. Δεύτερη ερώτηση. Όσον αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό, το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε τη στιγμή που βλέπουμε ότι ήδη υπάρχουν πολύ σημαντικές και προχωρημένες επιπτώσεις από τις ουσίες αυτές, ουσίες τις οποίες δεν έχουμε καταφέρει να οριοθετήσουμε παρκώς και για τις οποίες θα πρέπει να γίνει μια ενδελεχής σημαντική μελέτη και θα πρέπει τα πορίσματα της μελέτης αυτής να έχουν και ισχύ αναδρομική. Τρίτον, Ποια είναι η δική σα αντίδραση όταν βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη τι δικέ σα γνωμοδοτήσει ε, όσον αφορά του ε, επικονιαστέ. Ε? Πρόκειται η ΕΦΣΑ να απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πιο αυστηρή στάση απέναντι στι ουσίε αυτέ. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Γουλ. Χαίρομαι που είστε ανάμεσά μας. και θα χαιρόμασταν αν ε, υπήρχε υπάρξει ανανέωση της ε, θητείας σας. Και το σημαντικό είναι η ε, επιστημονική σκοπιά των πραγμάτων. Συνεχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η πολιτική προσπαθεί να επηρεαστεί από την δημόσια γνώμη. Έχουμε τα fake news, και σε έναν τομέα που κανονικά θα πρέπει να προσεγγίζεται επιστημονικός. Ε, βλέπουμε ότι έχουν και αυτά μία θέση ξαφνικά ε, και προσπαθούν να δράσουν και να επηρεάσουν μέσω των ε, fake news είπε ο κύριος Χόισλινγκ για επιστήμονες του Facebook, ένας όρος που περιγράφει ακριβώς αυτήν την κατάσταση η επιστήμη είναι γνωστή ότι εργάζεται αναλυτικά και χρειάζεται χρόνο. Και εμεί στο Κοινοβούλιο πρέπει να εργαζόμαστε έτσι και το είπε και ο συνάδελφο κ. Λίζα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας δίνει αυτόν τον χρόνο και αναφέρομαι συγκεκριμένα ε, στον κανονισμό για τα τρόφιμα όπου δράλες ε, και η Επιτροπή είναι ο νομοθέτης που δεν είναι. Θα πρέπει λοιπόν να το τονίσουμε αυτό στην Επιτροπή ότι δεν γίνεται έτσι. Πιστεύω λοιπόν ότι εμείς ε, ως ε, κομμάτι ε, του Ευρωπαίου νομοθέτη χρειαζόμαστε χρόνο για τόσο πολύπλοκα και τεχνικά θέματα. Θα πρέπει να εργαστούμε με λεπτομέρεια Ε, από την εμπειρία μου έχω προσέξει ότι πολλοί φάκελοι δεν συνάδουν με την πραγματικότητα, οπότε χρειαζόμαστε χρόνο φυσικά. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Χόισλινγκ όμως ότι η εναλλακτική ε, γεωργία δεν μπορεί να θρέψει ε, την, τον πλανήτη και ότι με αυτόν τον τρόπο εκπροσωπεί την βιομηχανία. τη βιομηχανία. Διαφωνώ με αυτό. Η εναλλακτική γεωργία χρειάζεται 6 ε, με 7 ε, φορές με μεγαλύτερη έκταση σε σχέση ε, με τους συνηθισμένους τρόπους γεωργίας. Αυτό το ξέρουμε αγαπητοί συνάδελφε. Και επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό ίσως θα ήταν και εναλλακτική για την εναλλακτική γεωργία η συμβατική γεωργία έχει και αυτές τις, ε, τους ε, υποστηρικτές της. Ε, θα έλεγα λοιπόν η πράσινη της Γερμανίας συγκεκριμένα να γίνει πιο θετική απέναντι στα γενετικά τροποποιημένα διότι έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούμε λιγότερα χημικά και λιγότερα μέσα όπως ε, για παράδειγμα εκλείονται ε, λιγότερες ποσότητες ε, διοξιδίου του άνθρακα. Μου ήταν σημαντικό λοιπόν να σας το υπενθυμίσω αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τον ε, κύριο Σκάνελ από την Επιτροπή που ε, θα ήθελα να πάρει το λόγο να απαντήσει τα όσα έχουν υποθεί, αν το επιθυμεί. Ε, thank you, Madam Chair. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι εδώ πέρα στα πλαίσια της παρουσίασης που έκανε ο κύριος Ούρλ όσον αφορά τον έπανα προσδιορισμό του στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της ΕΦΣΑ, πρόταση την οποία υποστηρίζει σαφώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΕΦΣΑ γνωρίζει την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα είναι δική σα σειρά εδώ στο Κοινοβούλιο να δείτε τις βασικές θέσεις του κυρίου Ούρλα. Είπε ο κύριο Ούρλα ότι θα ήθελε περισσότερο, μεγαλύτερο προπολογισμό για την ΕΦΣΑ, καλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την επιστημονική αξιολόγηση, πράγμα το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόταση που είχε υποβάλει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχει προσπαθήσει να υποστηρίξει ακόμα περισσότερο, όπου επιφέρουμε πολύ σημαντικέ αλλαγέ στην υφιστάμενη Γενική Νομοθεσία για τα τρόφιμα, αλλαγέ που θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΦΣΑ να έχει και του πόρου, αλλά και την νομική ικανότητα για να επιτύχει μεγαλύτερη διαφάνεια στα απορίσματα τα οποία προβάλλει προς τα έξω προς τους Ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά τα τρόφιμα. Εναπόκειται λοιπόν τώρα στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να νομοθετήσουν. Ξέρουμε ότι εσεί εκπονείτε μία έκθεση για το ζήτημα αυτό και η συγγήτρια μα έχει πει πάρα πολλέ φορέ εδώ στο Κοινοβούλιο ότι ήταν ε, δυσαρεστημένη με τον πολύ εσπευσμένο τρόπο με τον οποίο προωθείται η τροποποίηση αυτή τη νομοθεσία και ότι δεν δινόταν απαραίτητο χρόνο στο Κοινοβούλιο για να επεξεργαστεί την πρόταση αυτή. Εμεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίναμε συνεχώ εξηγήσει σε εσά και Ιδίω ο Επίτροπος Ανδρουκάητης αλλά και πρόεδρος Επιτροπής Γιούνκερ δώσανε πολύ μεγάλη σημασία στην πρόταση αυτή θέλοντας να δώσουν πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία στους πολίτες ότι όντως τους ακούμε, ότι τους αφογκραζόμαστε και ότι θέλουμε να αναλάβουμε σχετική δράση και μάλιστα με τρόπο αποφασιστικό και γρήγορο. Και για αυτό το λόγο σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αρχική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι τον Απρίλιο του 2018 μέσα σε τέσσερις μήνες δηλαδή καταφέραμε να υποβάλουμε μια πολύ φιλόδοξη πρόταση με τους απαραίτητους νοδευτικούς πόρου. Εμεί λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρήκαμε το χρόνο και την ενέργεια για να κάνουμε κάθε τι το αναγκαίο για να προωθήσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Και Εκτιμούμε αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να βρουν την απαραίτητη ενέργεια και του απαραίτητου πόρου για να ανταποκριθούν σε ένα σύντομο πιεσμένο χρονικό διάστημα. Και αποδεχτήκαμε επίση ότι ιδανικά θα έπρεπε να είχαμε περισσότερο χρόνο, αλλά προφανώ θα πρέπει να τηρήσουμε το κοινοβουλευτικό χρονοδιάγραμμα και παράλληλα θα πρέπει να παραμείνουμε φιλόδοξοι. Το επαναλαμβάνω αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόταση αυτή, όπω είπε και ο κύριο Ούρλα. Χρειαζόμαστε πραγματικά την απαραίτητη πολιτική βούληση για να προωθηθεί η πρόταση αυτή. Πρέπει να προσδώσουμε του απαραίτητου πόρου στην ΕΦΣΑ και θα ζητούσαμε και από τα άλλα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν την ηρωική αυτή προσπάθεια και να προχωρήσουμε γρήγορα. Γιατί θα είναι τεράστιο το επίτευγμα το οποίο θα καταφέρουμε να πετύχουμε εξ ονόματο θεσμικών μα οργάνων, αν από συλλογική πλευρά μπορούμε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να εγκρίνουμε μια σημαντικότατη απόφαση για να προσδώσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στο σημαντικότατο αυτό τομέα. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Εκτιμούμε την συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Τζόμερ, θέλετε να πάρετε το λόγο πάλι για να αντιδράσετε σε αυτά που ακούσαμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα πρέπει να απαντήσω σε αυτά που μόλις υποθέκαν ο εκπρόσωπος της ε, Επιτροπής ε, υπονοεί ε, ότι το κοινοβούλιο δεν είναι αρκετά φιλόδοξο, όπως επίσης και η συγγήτρια. Είναι ανοησία αυτό απαράδεκτο το γεγονός ότι η Επιτροπή μέσα σε μερικές, μερικούς μήνες ε, έκανε ε, την συγκεκριμένη πρόταση. Ε, ναι, όμως δεν υπάρχει αξιολόγηση αντικτύπου. και αυτό είναι το πρόβλημά μας και για το Συμβούλιο πρόβλημα. δεν υπάρχει αξιολόγηση αντικτύπου, το οποίο θα έπρεπε να είχε κάνει η Επιτροπή. Ε, και γι' αυτό το λόγο έχουμε τόσα μεγάλα προβλήματα το ότι θα πρέπει να δράσουμε με αυτή τη βιασύνη. Όταν λοιπόν δεν έχουμε τη δυνατότητα επαρκώς να συζητήσουμε με όλες τις, ε, με όλες τις πλευρές και με τις ΜΚΟ, τότε ε, δυσχεραίνεται το έργο μας ακόμα πιο πολύ και δεν εργαζόμαστε μονάχα πάνω σε ένα φάκελο και βρίσκω ενδιαφέρον επίσης το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει χρόνο και πόρους ε, διότι ε, συνηθίζει να λέει δεν έχουμε καθόλου ε, πόρους, καθόλου πόρους. Πολλά έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, όμως έχουμε την αίσθηση ότι δεν γίνεται τίποτα. Όσον αφορά την ε, φάκελο και τον κανονισμό ε, για την ε, πληροφόρηση περί των τροφίμων και εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ε, κανόνες και θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτή η αύξηση της διαφάνειας στην ΕΦΣΑ και η ΕΦΣΑ ε, θα έχει τα αναγκαία ε, χρηματοδοτικά κονδύλια και ότι θα συμμετέχουν και τα κράτη-μέλη. Όμως ε, δεν θέλω να μείνει έτσι ότι θα έρχεται η Επιτροπή και να λέει ότι η Επιτροπή είναι ο μόνος που ενδιαφέρεται για το καλό των πολιτών και ότι λαμβάνει σοβαρά τι ανησυχίε των πολιτών σχετικά με τον ε, με την γλυφοσάτη. όλοι θέλουμε διαφάνεια, θα πρέπει να γίνει ε, σωστά όμως. Έχουμε την ημερήσια διάταξή μα και η ημερήσια διάταξή μα λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει η πρώτη και η δεύτερη ανάγνωση, οπότε το θεωρώ ε, απαράδεκτο το πόσο ο επίτροπο παίρνει τηλέφωνα και προσπαθεί να επηρεάσει τους πάντες και να μην τηρήσει τον κανονισμό αλλά να υπάρξει μια επιταχυμένη διαδικασία που να περάσει από την πρώτη ανάγνωση. Σε μια τέτοια κατάσταση λοιπόν η Επιτροπή ε, περνά το 90% των προτάσεών της ε, και με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται ε, να περαστεί η πρόταση της Επιτροπής. Θέλουμε να ακολουθεί ε, η κανονική διαδικασία με πρώτη και δεύτερη ανάγνωση. Έπρεπε να το τονίσω αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Σόμα Λοιπόν, πολλά σχόλια έγιναν λέει η Πρόεδρος. Έχετε το λόγο αν θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, για την εμπιστοσύνη σας. Θα επανέλθω και στον κύριο Χόισλινγκ που εξέφερε μια επιφύλαξη για την εμπιστοσύνη. Για το περιεχόμενο η προτεραιότητα της δουλειά μας, η βάση της δουλειά μας είναι, ήταν και θα είναι η ποιότητα των επιστημονικών συμβουλών. Αν δεν το έχουμε αυτό, δεν πρέπει να επικοινωνούμε τίποτε. Θα πρέπει η ανάλυση επιστημονική να είναι ορθή. Και υπάρχουν διάφορες προκλήσεις μεθοδολογικές και άλλες και αυτό είναι το καθημερινό μας, ε, η καθημερινή μας δουλειά. Ο ΕΣΑ χρειάζεται τους πόρους από την άλλη μεριά για να παρακολουθεί τις καινοτομίε στην βιομηχανία των τροφίμων. Αν εμείς οι αξιολογητές κινδύνου δεν είμαστε ευθυγραμμισμένοι με την ταχύτητα του κλάδου του βιομηχανικού, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον, αν σκεφτείτε τα νανοηλικά ή τις χημικές ενώσεις τις οποίες είμαστε εκτεθειμένοι. Επομένως, το σημείο εκκίνησης πάντοτε πρέπει να είναι η πληρέστατη επιστημονική ανάλυση. Η άλλη, ε, το άλλο σκέλος είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πάντοτε ευθυγαμισμένοι με την κοινωνία και αυτό το πετυχαίνουμε και εδώ από εδώ στο σχόλιο το δικό σας. Όχι, δεν το καταφέραμε πάντοτε. Πρέπει να είμαστε σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς, με τις ε, ε, επιστημονικές πηγές και όλα αυτά προτού πάμε σε πολιτική σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Δεν έχουμε όμως κάποια μαγική λύση. Απλώς λέμε ότι η διαφάνεια δεν υπάρχει πλέον. Χρειαζόμαστε απόλυτη δέσμευση και συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, ώστε η κοινωνία των πολιτών να είναι, αν θέλετε, υπό κάποια έννοια συνυπεύθυνη των συστάσεων των δικών μας και των πορισμάτων μας. Να μην μιλούμε απλώς μια ψυχρή τεχνοκρατική γλώσσα, δηλαδή χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τις ανησυχίες των πολιτών. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, μόνο επιστημονική ανάλυση μπορούμε να κάνουμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω προς την κατεύθυνση της κοινωνίας των πολιτών. Τώρα τρίτον, πρέπει να χρησιμοποιούμε τις καινοτομίες της τεχνολογίας της ψηφιακής, των δεδομένων, του artificial intelligence, όλα αυτά δεν μπορούμε παρά μόνο να τα πετύχουμε σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να έχουμε ένα κόμβο που να είναι σε θέση να αναλύει την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία προτού αυτή ε, ε, διαδοθεί. Εάν δεν συνεργαστούμε με άλλους λοιπόν φορείς, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο έργο μας. Αλλά ποτέ καμία προσπάθεια δεν είναι επαρκής. Πάντοτε πρέπει να συνεργαζόμαστε περισσότερο με τους φορείς ε, τους υπεύθυνου για την, ε, τον έλεγχο των νόσων, τα χημικά εργαστήρια. Η συνεχιζόμενη συνεργασία, όπως έλεγα πριν, λοιπόν, είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας. Για τον κύριο Μπότς, κάναμε λάθη. Ναι, κάναμε λάθη. Προφανώς κάναμε λάθη, λέει ο μιλητής. και μάλλον υποτιμήσαμε τη συζήτηση για τον glyphosate. Οι επιστημονικές ενδείξεις επιβεβαιώθηκαν από όλες τις υπηρεσίες στον κόσμο με μόνη εξαίρεση το IRC του ΠΟΕ. Του ΠΟΕ με συγχωρείτε. Όλοι οι υπόλοιποι επιστημονικοί φορείς επιβεβαίωναν τις ενδείξεις που είχαμε, τις αναλύσεις που είχαμε. Επομένως, επιστημονικά σωστή ήταν η δουλειά. Σε επίπεδο επικοινωνία ήταν δύσκολο. Αλλά συχνά ακούμε από τους πολιτικούς, αν εσεί οι επιστήμονες κοινοποιούσατε καλύτερα, ενημερώνατε καλύτερα, θα διευκολύνετε και τη ζωή μας, τη δική μας δηλαδή, το δικό μας καθήκον. Όμω εμείς δεν μπορούμε να επικοινωνούμε, να κοινοποιούμε, να διαβιβάζουμε πολιτικές διαφορές. Αν υπάρχει πολιτική τάση ή διαφορά για το κατά πόσον πρέπει να χρησιμοποιούνται αγροχημικά ή όχι, αυτό δεν μπορεί να το επιλύσει η επιστήμη. Είναι πολιτικότατο ζήτημα για τις αξίες και το μέλλον της κοινωνίας μας. Άρα πρέπει αυτοί οι δύο κόσμοι να διαφοροποιηθούν. Να υπάρχει μια επιστημονική συζήτηση και μόνο μετά από αυτό μια πολιτική συζήτηση που δεν είναι δικό μας, ε, δική μας αρμοδιότητα βεβαίω. Έχουμε νομοθεσία για τα βιοκτώνα και ζανιοκτώνα έχουν αυτά κατανεμηθεί στους δύο οργανισμούς που έχουν κατανεμηθεί. Αν είναι σωστό, δεν ξέρω. Αυτό από εσά εξαρτάται. Εμείς συνεργαζόμαστε με τον ΕΚΤΑ σχετικά με, τους, ε, με τα στοιχεία σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταρακτές. σε πάση ο νομοθέτης αποφάσισε να διακρίνει τα βιοκτώνα και παραστοκτώνα σε δύο οργανισμούς. Εμείς ε, ρωτήσατε αν θέλουμε να είμαστε πιο γρήγοροι ή πιο καλοί. Εγώ θα σας δώσω την ε, προκλητική απάντηση που θέλουμε να είμαστε γρήγοροι και καλοί. Λέτε ότι είναι ευθυνή απάντηση τώρα. Ε, εγώ απλώς υπογραμμίζω τη δική μας θέση. Εσείς είσαστε οι νομοθέτες τέσσερα μέλη του Κοινοβουλίου μας οδήγησαν στο δικαστήριο. Επειδή δεν αποκαλύπταμε τις πηγές, τις πληροφορίες που μας ζητούσαν στην περίπτωση glyphosate. Και είμαστε στο δικαστήριο, που δεν είναι και θαυμάσιο. Να οδηγεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον ΕΦΣΑ στο δικαστήριο δεν είναι ιδανικό. Θα ήμασταν απόλυτα ικανοποιημένοι με ένα σαφ σαφέ νομοθετικό πλαίσιο με το μέγιστο επίπεδο της ε, διαφάνειας καταλαβαίνοντας ότι υπάρχουν ε, θέματα ε, διανοητικής ιδιοκτησίας ώστε να μπορέσουμε αυτή τη διαφάνεια να την, να την υλοποιήσουμε, να την κάνουμε πραγματικότητα. Και αν τώρα αναβληθεί το θέμα, καταλαβαίνω τα επιχειρήματα της κυρία Ζώμα, αλλά αν αναβληθεί, τότε πάλι ο ΕΦΣΑ θα την πληρώσει υπό την έννοια της εικόνας και της αξιοπιστίας, γιατί πάλι εμάς θα κατηγορούν ότι δεν είμαστε διαφανείς. Επομένως, για εμάς και για τους πολίτες είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, όμως λυπάμαι, εγώ δεν μπορώ να σας επιβάλλω κάτι, εμείς θα αποδεχθούμε οτιδήποτε αποφασίσετε, είναι δική σας η απόφαση. Αν θέλετε να το αναβάλλετε, θα ακολουθήσουμε. Απλώς λέω ότι έχουμε κάθε συμφέρον στην ταχύτερη δυνατή απόφαση επ' αυτού. Αλλιώς θα υπήρχε, θα υπήρχε κάποια αντίφαση. Εκτός μικροφώνου κάτι λέει. Καταλαβαίνω και αποδέχομαι αυτό το οποίο λέτε. Ενδεχομένως να μην χρησιμοποίησα σωστά τον όρο αναβολή και μετάθεση. Απλώς δημιουργήθηκε μία αναμονή από τη δική μου την πλευρά ότι ενδεχομένω να μπορούσαμε να προχωρούσαμε λίγο πιο γρήγορα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά από ό,τι φαίνεται εσεί δεν προτίθεστε να προχωρήσετε πάρα πολύ γρήγορα με τη μεταρρύθμιση τη Γενική Νομοθεσία για τα τρόφιμα. Κατά αυτόν τον τρόπο χρησιμοποίησα τον όρο αναβολή. Κυρία Μάισνερ, αναφερθήκατε στο ζήτημα τη επικοινωνία και θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα προκειμένου. Όσον αφορά την μικροβιακή ανθεκτικότητα, νομίζω ότι εδώ η ανακοίνωσή μας είναι πολύ καλή και με το ECDC και με την Ευρωπαϊκή Αρχή για τα Φάρμακα. Δεν θα έλεγα την αδύναμη λοιπόν η στάση μα, και θέσατε ένα σημαντικό ερώτημα. Πόσα χρήματα θα χρειαστεί η ΕΦΣΑ. Θα συνέκρινε εδώ πέρα την ΕΦΣΑ με την Ευρωπαϊκή Αρχή Φαρμάκων. Ουσιαστικά αυτοί έχουν το διπλάσιο προσωπικό, εμεί έχουμε 500 και αυτοί 1000 άτομα, αλλά έχουν τέσσερι φορέ τετραπλάσιο προπολογισμό σε σχέση με εμά. 350 περίπου εκατομμύρια έχουν για φέτος, εμεί μόνο 80. Μα μόνο και μόνο αυτό τα λέει όλα. Γι' αυτό το λόγο αίμα μπορεί να λειτουργήσει τελείω διαφορετικά με του πυρογνώμονε. Γιατί μπορούν πραγματικά να πληρώσουν τι αρμόδιε αρχέ στα κράτη-μέλη για να του δανείσουν εντό ε, εισαγωγικών του εμπειρογνώμονε. Εμείς δίνουμε μόνο 7,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ποσό το οποίο δίνει αίμα είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερο. Θα ήταν ε, πάρα πολύ καλό να μπορούσαμε να είχαμε ένα προπολογισμό των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα είχαμε μία εύσα η οποία θα ήταν σε απόλυτη ετοιμότητα, θα μπορούσε πραγματικά επιστημονικά να παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις στον τομέα των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και το καθεξής. 200 λοιπόν εκατομμύρια θα ήταν ένα τιτανικός προπολογισμός για μας, ετήσιος βέβαια. Κύριε Χάουσλινγκ, λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη τα όσα είπατε δεν μπορεί να είναι ποτέ βέβαια πολιτικό ο δικό μου ρόλο και ξέρω ότι μερικέ φορέ φτάνω λίγο στα άκρα. Λόγω τη φύση μου συμβαίνει αυτό, σα ζητώ συγγνώμη. Παρ' όλα αυτά, λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη τα όσα μου υπενθυμίσατε. Μου είπατε ότι εκπροσωπώ μια επιστημονική οργάνωση. Το λαμβάνω αυτό σοβαρά υπόψη, σαφώ. Και ενδεχομένω να είμαι όντω πιο προσεκτικό στο μέλλον. Τα όσα είπατε όμω σε σχέση με τη συνέντευξη που έδωσα σε μια αυστριακή εφημερίδα πρόσφατα, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε κατηδίων λίγο περισσότερο στα γερμανικά. Είπα ότι ε, η βιολογική γεωργία είναι πολύ σημαντική, αλλά είπα ότι χρειαζόμαστε μια εντατική κυκλική και βιώσιμη γεωργία, προκειμένου να καταφέρουμε να θρέψουμε 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Και όσον αφορά την γονιδιακή τεχνολογία, δεν είπα ότι θα προωθούσα σών και καλά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, είπε ότι θα πρέπει να καλύψουμε τις ζημίες που υπάρχουν πριν και μετά τις συγκομιδής στις αναπτυσσόμενες χώρες και έπειτα θα αναφερόμουν ενδεχομένως την πιθανή χρήση των προϊόντων αυτών στον προηγμένο κόσμο. Και μόνο τότε πραγματικά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ειλικρινά για το αν μπορεί να βοηθήσει ή όχι η γονιδιακή τεχνολογία. Και για το ζήτημα μας αυτό, από επιστημονικής πλευράς, κάνουμε τις απαραίτητες αναλύσεις. Θα ολοκληρώσω το σημείο αυτό και κάτι ακόμα, αν μου το επιτρέπετε. Μα ρωτήσατε αν απομακρυνόμαστε από την αρχή τη προφύλαξη. Μα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφεί. Η επιστήμη δεν χρησιμοποιεί αρχή προφύλαξη. Εμεί κάνουμε ανάλυση κινδύνου. Εσεί μετά ω πολιτικοί παίρνετε τα δικά μα επιστημονικά δεδομένα και χρησιμοποιείτε και άλλου θεμητούς παράγοντες όπως οικονομική μεγέθυνση, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές κτλ. Και εσείς αποφασίζετε ως ηθήνοντες χάραξης πολιτικής για το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι η αρχή της προφύλαξης. Οι επιστήμονες δεν μπορούν να αποφασίσουν για την αρχή της προφύλαξης. Οι επιστήμονες παράγουν επιστημονικά δεδομένα. Εσείς τα χρησιμοποιείτε και τα συνδυάζετε με άλλα δεδομένα και αποφασίζετε για την αρχή της προφύλαξης. Μόνο εσείς. Κυρία Μελιόρο, τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε, μας ρωτήσατε, προκειμένου να τροφοδοτήσουμε λίγο περισσότερο μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους εμπερογνώμονες των κρατών μελών. Στα πλαίσια του πυλώνα βιωσιμότητας επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει πει ότι ε, θα μπορούσαμε να τονώσουμε λίγο περισσότερο τους οργανισμούς αυτούς οι οποίοι απασχολούν τους εμπειρογνώμονες προκειμένου να έχουν, ε, αν θέλετε, να είναι πιο διαθέσιμοι να μα δανείσουν αυτού του εμπειρογνώμονε, αν εμεί μπορούμε να του δίνουμε μία αμοιβή, αν μπορεί να γίνεται αυτό μεταπληρωμή. Αυτό θα μείωνε κάπω την πίεση, μείωση, την πίεση, με συγχωρείτε, προ τι αρμόδιε εθνικέ αρχέ, οι οποίε μα λένε ότι σαφώ θα θέλαμε να σα δώσουμε εμπειρογνώμονε, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί του χρειαζόμαστε εδώ, στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι όντω αν υπήρχε το κίνητρο αυτό το οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λυνόταν το πρόβλημα αυτό. Επίσης, οι εμπειρογνώμονες είναι πλέον επιστημονική συγγραφή όσον αφορά τα άρθρα τα οποία δημοσιεύουμε. Δύο εκατομμύρια downloads είχαμε πέρυσι για τις επιστημονικές γνώμες, τα επιστημονικά άρθρα μέσω του επιστημονικού περιοδικού της ΕΦΣΑ. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Χρειαζόμαστε όμως μια πολιτική δήλωση από τα κράτη-μέλη που να λέει ξεκάθαρα ότι θέλουν να συνεχίσουν να προωθούν το ευρωπαϊκό σχέδιο όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Χρειάζεται και μια πολιτική δήλωση. Καταλαβαίνετε ότι είναι διτό το σχέδιο αυτό. Προφανώς τα κράτη-μέλη παρέχουν επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν δεν υπάρχει το απαραίτητο χρηματοδοτικό σύστημα, τότε δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την εργασία αυτή η μεγαλύτερη απειλή είναι να μην έχουμε του απαραίτητου εμπειρογνώμονε, επειδή θα διστάσουν να μα του παράσχουν οι αρμόδιε αρχέ των κρατών μελών. Το χρονοδιάγραμμα για τη Γενική Νομοθεσία για τα Τρόφιμα νομίζω ότι το συζητήσαμε εκτενώ με τα υπόλοιπα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ετέθησαν κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση, τη σύγκρουση συμφερόντων, τη διαφάνεια. Νομίζω ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στο ζήτημα τη διαφάνεια. Μα δίνει κάποια ε, δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν εκ των προτέρων να κοινοποιούνται. Προβλέπετε μια συγκεκριμένη συνεργασία με τους υπερογνώμονες της ΕΦΣΑ. Αναφερθήκατε στους ενδοκρινικούς διαταρακτές. Σαφώς το ζήτημα αυτό μας απασχολεί και εμάς στην ΕΦΣΑ, στο ζήτημα των, στον τομέα των ζυζανιοκτώνων, στον τομέα των πρόστων των τροφίμων και προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στην επιστημονική βιβλιογραφία για να έχουμε την καλύτερη δυνατή επιστημονική ανάλυση όσον αφορά τις ουσίες αυτές. Θα πρέπει να γνωρίσουμε όμως ότι εδώ πάλι το νομικό πλαίσιο με την ΕΚΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Ουσιών και το νομικό πλαίσιο που έχει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων δεν είναι ευθυγραμμισμένα. Επομένω και αυτό δημιουργεί κινδύνους. Για ποιο λόγο τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ακολουθεί τις γνωμοδοτήσεις της ΕΦΣΑ Μα κοιτάξτε, αυτό είναι δικαίωμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σαφώ μπορούν να συμβουλεύονται τη δική μα την επιστημονική γνωμοδότηση, αλλά μπορούν να λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα δεδομένα. Εμεί έχουμε καθαρά συμβουλευτικό ρόλο. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τη δική μα την επιστημονική γνωμοδότηση. Μόνο αυτοί οι οποίοι νομιμοποιούνται πολιτικά και δημοκρατικά μπορούν να πάρουν πολιτικέ αποφάσει για την κοινωνία, όχι εμεί ω επιστήμονε στα πλαίσια τη ΕΦΣΑ. Τούτων λεχθέντων ολοκληρώνω την εισήγησή μου. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντόρφαν, θέλετε να πάρετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Ουόλ, θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, για νέα ε, ζυζάνια τα οποία ε, καταφτάνουν στην Ευρώπη διότι είμαστε συνδεδεμένοι με το διεθνές εμπόριο. Έχουμε διάφορα τέτοια Ε, δεν έχουμε στην Ευρώπη ακόμα τα απαραίτητα ζεζανοϊκτώνα για να τα αντιμετωπίσουμε ε, και ε, θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 350 να, κάνουμε, να έχουμε παρεκκλήσεις το οποίο οδηγεί σε κριτική Ε, γνωρίζετε το πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε, να το επιταχύνουμε, ούτως ώστε να αντιδράσουμε σε αυτές τις προκλήσεις και δεύτερον, πολύ συχνά στις χώρες προέλευσης αυτών των ζημιοκτώνων υπάρχουν ε, υπάρχουν άλλα ζυζάνια τα οποία τα καταπολεμούν, όμως θα μπορούσαμε ίσως να τα εισάγουμε όμως υπάρχουν ε, περιορισμοί, δεν μπορούμε να εισάγουμε ε, κάτι τέτοιο από το εσωτερικό, πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε ώστε να υπάρχει μια βιολογική καταπολέμηση τέτοιων ε, ζητανίων. Και ο κύριος Χάουσλινγκ. Ευχαριστώ και πάλι. το Facebook Science ε, δεν είναι σαν να λέμε εμείς είμαστε οι καλοί και οι άλλοι όχι ε, και στον κύριο Πορτιέ ε, είστε επιστήμονας όμως έχουν βγει που έδειξαν το αντίθετο λέτε δηλαδή λες και μονάχα εσείς έχετε δίκιο και όλοι οι άλλοι άδικο στα νεονικοτινοειδή για παράδειγμα ε, είχε υποθεί πριν κάποια χρόνια ότι δεν δημιουργούν ε, προβλήματα. Η κυρία Ζώμα φεύγει, όμως ε, είπε για τους αριθμούς ότι για την εναλλακτική γεωργία χρειαζόμαστε 6 με 7 φορές μεγαλύτερες εκτάσεις. Δεν ξέρω πού βρίσκεται τέτοιους αριθμούς. θα πρέπει να ξέρετε ότι και με τη χημεία έχουμε προβλήματα. 70% ε, λιγότερα ε, εντομοκτώνα και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε έτσι ξαφνικά όλα είναι υπέροχα και ωραία. Μπορούμε να το συζητήσουμε μεταξύ μας. Άμα θα μπορούσατε όμως να απαντήσετε σε αυτό, παρακαλώ. Έχετε το λόγο, λέει η Πρόεδρος. Ε, κύριε Ντόφμαν, δύσκολες οι ερωτήσεις σας και αφορούν εις τους διαχειριστές κινδύνου ε, για τους ανταγωνιστές ε, ε, παρασίτων των φυτών. Αυτό δεν είναι θέμα του ΕΦΣΑ. Ίσως μπορούμε να συζητήσουμε διμερώς για το τι μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτό. Τώρα για το άρθρο 3-3. Αυτό ξέρετε από τα κράτη-μέλη πρέπει να πω. κατά πόσον δηλαδή μπορεί κανείς να παρεκκλίνει με εξιωτήσεις ε, επίγουσες για νεοαναδιόμενα παράσιτα και εδώ δεν μπορώ να συνεισφέρω ιδιαίτερα γιατί δεν εμπίπτει στην εντολή του ΕΦΣΑ. Στο σημείο που σας απογοητεύω. Εμείς ασχολούμαστε με τις δραστικές ουσίες, τα MRL, αλλά όχι την ε, διαχείριση κινδύνου των ε, προϊόντων προστασίας των φυτών. Ε, και κύριε Χόισλινγκ, με χαρά να επανέλθω, αλλά πρέπει να είμαι συγκεκριμένος και έχει καταγραφεί 1η Δεκεμβρίου του 2015 τα όσα είχα πει εάν οι επικριτές η ΕΦΣΑ αποστείλουν επιστολή υπογεγραμμένη από 96 επιστήμονες σχετικά με σφάλματα που έχουμε κάνει, μία εβδομάδα μετά την δημοσίευση 5.000 σελίδων και άνω για το glyphosate, έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί να είχαν επαρκή χρόνο εντός μίας εβδομάδας να διαβάσουν αυτές τις 5.000 σελίδες και επομένως αυτή ήταν η άποψη που είχαν ήδη πριν δημοσιευθούν αυτά τα έγγραφα. Αυτό είχα πει. Αν λοιπόν η επιστήμη ε, είναι βρεθεί μάλλον στο πεδίο της ε, διαφοράς απόψεων, τότε μου θυμίζει το Facebook και τη δική του επιστήμη. Γιατί είναι αξίες αυτά, μεταλλασσόμενες. Είναι εκστρατεία πολιτική. Δεν είναι επιστήμη. Και τότε ας μην του δίνουμε το μανδύα του επιστημονικού. Ας πούμε, δεν το θέλουμε, κάνουμε μια εκστρατεία εναντίον του, αλλά ας μην λέμε ότι αυτά βασίζονται σε επιστημονικές ενδείξεις. Είναι θέμα ψήφων. Υπέρ, κατά. Ξανά παραπέμπω στην επιστήμη του Facebook. Επιστήμη εντός οικών. Πάντως ε, ε, καταγράφει το τι είπα και είναι σαφές. Ο κύριος ε, Ποχτιέ είναι εξαιρετικός επιστήμων και δεν θα τον επέκρινα ποτέ, δεν θα υπέσκαπτα ποτέ την αξιοπιστία του. Αλλά ο, Παχ... κύριος Ποχτιέ επίσης είναι σύμβουλος δικηγορικών γραφείων στις Ηνωμένες Πολιτείες που ασχολούνται με συγκεκριμένες δικαστικές διαφορές έχει συγκεκριμένα συμφέροντα και εσείς είστε οι πρώτοι που ζητάτε τα συμφέροντα αυτά να είναι διαφανή. Το ζητάτε από εμά, από τον ΕΦΣΑ. Επομένως, η κάθε άποψη πρέπει να ε, ερμηνεύεται σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί δεν πρέπει να θεωρούμε ότι εμείς είμαστε καλοί και οι άλλοι είναι οι κακοί και εάν αυτή είναι η εντύπωση που δίνουμε πρέπει να την αλλάξουμε. πρέπει να είμαστε ταπεινοί διότι γνωρίζουμε με βάση την, τα επιστημονικά προηγούμενα ότι αυτό που θεωρούμε ότι γνωρίζουμε σήμερα μπορεί αύριο να αποδειχθεί εσφαλμένο. Βεβαίως, από την άλλη, πρέπει να επιμένουμε σε αυτό που είναι γνωστό σε μας επί τη βάση της επιστημονικής ένδειξης. Αν όμως δίνουμε την εντύπωση Τη υπεροψία ότι εμείς ξέρουμε καλύτερα από τους άλλους, τότε αυτό σίγουρα πρέπει να το αλλάξουμε. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ τον δόκτορα Ουόλ. Μετά από την σημερινή συνάντηση θα ακολουθήσουμε βεβαίως τη διαδικασία και θα, θα μάθετε βεβαίως το πόρισμα. Ευχαριστώ όλους. Αυτά, εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή συνεδρίαση. Καλό γεύμα σε όλους.